Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζουμε τη συνεδρίασή μα. Αν δεν υπάρχει καμιά πρόταση για αλλαγέ στην ημερήσια διάταξη, αυτή εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο, έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίασεώς μα στις 11 η Μαΐου. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, εγκρίνονται και τα πρακτικά αυτά. Επόμενο θέμα. Ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Δεν έχω ανακοινώσει σήμερα, οπότε περνάμε ευθύ αμέσω στην ακρόασή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα η ακρόασή μας έχει να κάνει με την ισότητα των φίλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να καλωσορίσω εδώ όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως τους προσκεκλημένους μας εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ακράση αυτής. Πρόκειται για την ε, πλατφόρμα που το 95 που ήδη αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η σχέση των μέσων ενημέρωσης με τις γυναίκες. Η συμμετοχή των γυναικών σε υψηλές θέσεις στα μέσα ενημέρωσης παραμένει πάρα πολύ χαμηλή. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι γίνεται με την επικοινωνία υψηλού επίπεδου και πώς τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να συνεισφέρουν στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η δημόσια αυτή ακρόαση θα εξετάσει πώς η παρουσία των γυναικών στη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης αλλά και στις θέσεις αποφάσεων που λαμβάνονται υποφάσεις δηλαδή στα μέσα ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της νοοτροπίας υπέρ της ισότητας. Πώς θα καταπολεμηθούν τα στερεότυπα στα μέσα ενημέρωση σε βάρος των γυναικών, όπω επίση και οι τάσει, αλλά και οι αλλαγέ που παρατηρούνται στις δομέ που έχουν να κάνουν με την ισότητα στα μέσα ενημέρωση. Θα ακούσουμε και από τον ίδιο τον κλάδο αλλά και από τους χρήστες και θα δούμε πώς αυτοί οι δύο παράγοντες αλληλεπιδρούν ένα στον άλλον. Έτσι θα συλλέξουμε πολύτιμες πληροφορίες εν ώψη της έκθεσης που συντάσσουμε με τον ίδιο τίτλο. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μιχαήλα Σόντροβα από την Επιτροπή μας, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Όμως μας στέλνει ένα μήνυμα βιντεοσκοπημένο, το οποίο και θα παίξουμε τώρα. Μήνυμα λοιπόν από την συγκέντρια. Παρακαλώ. Colleagues, I am sending my warmest greetings from Prague. I for not being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 fruitful discussion and I hope uh, see you later, see you soon in Brussels. Dear colleagues, I am sending Thank you very much. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ την Μικαέλα Σόντροβα για το βίντεο αυτό. Τώρα λοιπόν θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, στους ειδικού που έχουμε εδώ μαζί μας. Και πρώτα απ' όλα στην κυρία Λέγκα Βοτσόκοβα, που ασχολείται με τις κοινωνικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Charles Καρόλου, δηλαδή, στην Πράγα. Ε, Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την παρουσίαση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 παρουσιάσω τις θέσεις μου. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν ε, με μια πλήρη επισκόπηση των φεμινιστικών ε, θεωριών, των θε, θεωριών σχετικές με τη διάσταση του φύλου, με έναν ιδιαίτερο παράγοντα λοιπόν. Βλέπω ότι δεν μπορείτε να δείτε όμως τις διαφάνειες της ε, παρουσίασής μου. Επιπλέον υπάρχει φοβερό πρόβλημα σε σχέση με τον ήχο που βγαίνει από τα γερμανικά. Ε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα μικρόφωνα που χρησιμοποιούνται προς τα γερμανικά. Λοιπόν, οι μελέτες για, ε, για το φύλλο ασχολούνται με αυτή την προοπτική, με έρευνες και παρουσιάζουν νέα δεδομένα. Εάν μελετήσουμε τα μέσα, δεν μπορούμε να απομονώσουμε τον παράγοντα του φύλου από άλλες πτυχές κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές, βέβαια. που επηρεάζουν ε, τον ρόλο και τον τρόπο εργασίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τις δομές που ασχολούνται με την διάσταση της παραγωγής και των προϊόντων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι αυτοί οι τομείς δεν μπορούν όμως να εξεταστούν αποκομμένοι και τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ έντονη βέβαια η παρουσία τους ε, στα μέσα. Οι μελέτες ε, σχετικές με τα ΜΜΕ θα πρέπει να στηρίζονται βέβαια σε γεγονότα, ε, σε δεδομένα, τα οποία όμως είναι δύσκολο να συλλεγούν. Δεδομένα τα οποία σημαίνουν αξιολόγηση της επίδρασης που μπορεί να έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω της παραγωγής τους στην κοινωνία και την οικονομία γιατί μας ε, απαντούν πάντα τα ΜΜΕ ότι τα προϊόντα τους απευθύνονται απλώς στο κοινό τους, παράγονται για το κοινό τους. Και άρα παράγουν αυτό το οποίο ζητά, ζητεί το ακροατήριο, το κοινό. Αλλά ότι δεν καθοδηγούν το προϊόν. Τώρα, τι προκύπτει σε σχέση με τα γεγονότα, με τα στοιχεία οι μελέτες λοιπόν για τη θέση των φίλων στα ΜΜΕ κοιτούν και τη γυναίκα ως εργαζόμενη, ως δημοσιογράφο, ρεπόρτερ και το καθεξής. Αλλά παράλληλα από την τελευταία επισκόπηση των ΜΜΕ της σειράς ε, που διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια έγινε, είδαμε ότι έγινε η μελέτη με μία μόνο ημέρα έρευνας Άρα και η μεθοδολογία ήταν ε, περιορισμένων, ε, περιορισμένης εμβέλειας και δεν μπορεί να είναι επιστημονικά αξιόπιστη. Εδώ βλέπουμε στοιχεία λοιπόν που μας ε, παρουσιάζουν θέσεις των γυναικών σε 37, των, ε, των θεμάτων των σχετικών ε, με την, που παρουσιάζονται από γυναίκες στη συγκεκριμένη ημέρα της έρευνας στο 37% άρα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης η ηλικία έχει πολύ μεγάλη σημασία για την παρουσία της γυναίκας στην οθόνη. Όσο πιο ηλικιωμένη η γυναίκα, τόσο πιο περιορισμένες οι πιθανότητες να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης. Το περιεχόμενο σε όλο και πιο περιορισμένο βαθμό παράγεται από γυναίκες και έχουμε και την ε, οριζόντια ή εγκάρσια διαχωριστική γραμμή. Αυτά τα ε, αντικείμενα εργασία των ΜΜΕ που μπορούν να χαρακτηριστούν ως σκληρός πυρήνας ή ως πιο ε, ελαφρύ περιεχόμενο. Οι σοβαρές λεγόμενες ειδήσει ανήκουν στο πεδίο δραστηριότητας των ανδρών, ενώ οι πιο ελαφρές των γυναικών, κατά κύριο λόγο. Ένα μόνο τρίτο το εις θερματολογίας με το οποίο ασχολούνται γυναίκες δημοσιογράφοι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως σοβαρό περιεχόμενο. Διαχωρισμός επίσης σε σχέση με την ιεραρχία. Πόσες είναι οι γυναίκες που έχουν φτάσει σε ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας και εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πάντα το λεγόμενο η λεγόμενη η άλλη οροφή, ότι δηλαδή οι γυναίκες δεν μπορούν να φτάσουν σε ανώτερες ε, θέσεις διοικητικές. Αν και πάλι εδώ είναι δύσκολη συλλογή καλής ποιότητας δεδομένων ε, σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Πάντως τα στοιχεία που έχουμε από το 2011 μας δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι οι λιγότερες, είναι σημαντικά λιγότερες στις ε, ηγετικές θέσεις, στις διευθυντικές σχέσεις από ότι οι άντρες. Η θεματολογία επίσης που επιλέγεται σε σχέση με την ε, με το συγκερασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου βίου, θέματα harassment, παρενόχλησης δηλαδή ή άλλα κοινωνικής ε, παρενόχλησης όπως το λεγόμενο mobbing, σε ποιο βαθμό απασχολούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή η φαλοκρατική αντιμετώπιση των γυναικών όταν αυτές εργάζονται ως ε, δημοσιογράφοι. Εδώ βλέπουμε να εντείνονται αυτά τα φαινόμενα και μάλιστα ε, εντείνονται και οι επιθέσεις, οι λεγόμενες ad hominem, οι επιθέσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με την εξωτερική εμφάνιση, ε, αν είναι καλοντημένη, αν είναι όμορφη κτλ. μια γυναίκα. Αυτό βλέπουμε να πολλαπλησιάζεται και ιδιαίτερα λόγω των ε, κοινωνικών δικτύων. Οι προοπτικές επίσης, ε, οι τάσεις δηλαδή που μπορούμε να διαπιστώσουμε Και εδώ προσπαθούμε να κάνουμε μια επισκόπηση των δυνατοτήτων ε, για αλλαγές στο μέσο στα μας μαζικής ενημέρωσης συνολικά ως ε, κλάδο σε σχέση με τη θέση των γυναικών, το περιεχόμενο, το σχετικό με τις γυναίκες, αλλά και τα ποσοστά συμμετοχής ε, των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Και βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερη η εμφάνιση θεμάτων σχετικών με τις γυναίκες όταν και ο ρυθμός των εργαζομένων γυναικών είναι υψηλός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει λοιπόν διασύνδεση, σύνδεσμος μεταξύ του λεγόμενου περιεχομένου των γυναικών και, τον αριθμό των, και του αριθμού των γυναικών δημοσιογράφων. Δεν είναι αυτό νομίζω μια ευθεία σχέση. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε όσο πιο πολλέ είναι οι γυναίκες, τόσο πιο πολλά τα φεμινιστικά θέματα. Δεν είναι απαραίτητο αυτό να ισχύει. Ένα άλλο κλισέ που ακούγεται επίση είναι ότι όταν έχουμε γυναίκε σε ηγετικέ θέσει των μέσων μαζική ενημέρωση, αλλάζει σημαντικά το περιβάλλον ε, και το περιεχόμενο. Πάλι με τα δεδομένα που έχουμε στη θέση μα μπορούμε να διαψεύσουμε αυτή την δήλωση, δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Στον κλάδο των ΜΜΕ, όταν λαμβάνουν γυναίκες και βλέπουμε ότι έχουν την ίδια συμπεριφορά και τις επιλογές ε, με τους άντρες. Επίσης τώρα μια παράθεση του βιβλίου της κυρίας Βαν ε, για τη θέση των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας λέει ότι είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε τους τρόπους βελτίωσης της υποεκπροσώπησης, γιατί είναι πολύ σημαντική η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα ΜΜΕ. Ωστόσο αυτό, σημειώνουμε, δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση του περιεχομένου των ΜΜΕ. Και γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι συσχετισμοί, γιατί εμφανίζονται ως ψευδία σε αυτοί οι ισχυρισμοί που σας ανέφερα νωρίτερα. Πρώτον, διότι δεν είναι διαδική κατηγορία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή το περιεχόμενο δεν προσδιορίζεται μόνο ε, μεταξύ ανδρικής ή γυναικείας επιλογής. Δεν επιλέγει κανείς μια, ένα περιεχομένο μόνο επειδή είναι άντρας ή μόνο επειδή είναι γυναίκα. Επίσης, Μπορεί με να υπάρχουν κοινέ εμπειρίε σε σχέση με τι γυναίκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η επιλογή ενό άνδρα μια γυναίκα ε, στο ίδιο πόστο θα οδηγούσε σε περιεχόμενο διαφορετικό. Επίσης ε, η έννοια της ε, τυφλότητας ως προς το φύλλο. Πολύ συχνά σημειώνεται ότι οι γυναίκες που εργάζονται στα ΜΜΕ ε, είναι επιδεικνύουν τυφλότητα όπως υπήρουν ουδέτερες ως προς τα θέματα τα γυναικεία. Μπορεί αυτό βεβαίως ε, να ισχύει, αλλά ίσως ε, εξηγείται και από το γεγονός ότι η προβολή των γυναικείων χαρακτηριστικών ή του γυναικείου τύπου συνιστά αδυναμία και είναι προτιμότερη η επίδειξη ε, ανδροπρεπών χαρακτηριστικών και για την αναγνώριση της οποίας θα τύχει μια γυναίκα στο χώρο εργασίας. Ε, η αντίληψη επίσης ε, του ότι η συμμετοχή των γυναικών στα ΜΜΕ θα μπορούσε με την προβολή παραδείγματι των επαγγελματικών τους επιλογών να ε, οδηγεί σε μια αλλαγή επιλογών. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αν κάποιος ασχολείται με θέματα σχετικά με το φύλλο, υπερβολικά, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα δημοσιογράφος, επικρίνεται για μια υπερβολικά ιδεολογικά φορτισμένη επαγγελματική λογική. Δηλαδή ε, ε, βρίσκεται σε μειονεκτική ε, θέση. Ε, βλέπουμε ότι στα ΜΜΕ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της αντικειμενικότητας. Όλοι λένε «Α, πρέπει να είναι αντικειμενικές ειδήσει, αντικειμενικές ειδήσει και τίποτε άλλο». Σωστό είναι αυτό μεν. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν κάποιες πτυχές που έχουν να κάνουν με το αν είναι κανείς άντρας ή γυναίκα και που λόγω του φίλου τους μπορούν να οδηγήσουν διαφορετικά αποτελέσματα σε επιλογές περιεχομένου, ακόμα και σε πολιτικού περιεχομένου επιλογές. Άρα μπορεί η αντικειμενικότητα να είναι σημαντική, αλλά πολύ πιο σημαντική είναι η ουδετερότητα, η, ανεξαρτησία, η ανεξαρτησία περισσότερο, η ουδετερότητα από οποιαδήποτε πολιτική ε, επιρροή. Και βέβαια η οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία των ΜΜΕ έχει τεράστια σημασία. Βλέπουμε πολύ συχνά ότι τα ΜΜΕ είναι προσανατολισμένα στο οικονομικό κέρδος πάνω απ' όλα και ότι πολλές φορές κάποιες ε, δημοσιογραφικές ή άλλες επιλογές σχετικές με το περιεχόμενο των δημοσιογράφων έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις οικονομικές επιλογές των ε, ε, εργοδοτών τους, των ε, ιδιοκτητών των ΜΜΕ. Και εδώ περνάμε σε μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει με την ε, υπογράμμιση τις της γυναίκας στα, μέσα από τα ΜΜΕ. Μια παγίδα θα την χαρακτηρίσω. Από τη δεκαετία του 70 αλλά και του 80 ιδιαίτερω είδαμε να ενισχύεται ο γυναικείος πληθυσμό στα ΜΜΕ και γιατί βέβαια απευθύνονταν αυτά σε ένα πιο ποικίλο πληθυσμό με γυναίκες ε, ως κοινό και άρα θεωρήθηκε ότι είναι σκόπιμο να υπάρχουν και γυναίκες παρουσιάστρες εκπομπών αλλά και περισσότερες εκπομπές με περιεχόμενο lifestyle και άλλα τέτοια. Και τελικά προβλήθηκαν εικόνες και επιλογές οι οποίες οπωσδήποτε δεν ήταν ε, ισορροπημένες σε σχέση με την προσέγγιση των φίλων και την ισότιμη μεταχείριση. Και ναι λοιπόν μπορεί να υπήρχαν περισσότερες γυναίκες ε, στις εκπομπές, αλλά αυτές με την παρουσία τους και τη συμπεριφορά τους στις εκπομπές αυτές, απλώς ενίσχυαν τα στερεότυπα. Άλλη μία παγίδα λοιπόν. Και επίσης μια άλλη παγίδα που ήθελα να επισημάνω είναι ε, το θέμα της ηλικία, η παρουσία των ε, ηλικιωμένων γυναικών, πιο ηλικιωμένων γυναικών στα ΜΜΕ είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Όσο καλές και μάλιστα μπορούν να είναι πολύ καλές οι γυναίκες, εφόσον είναι πιο προχωρημένης ηλικία έχουν πολύ περιορισμένες ευκαιρίες για παρουσία στα ΜΜΕ. Αυτή είναι η παγίδα όπως τη χαρακτηρίζουμε. Το ίδιο βλέπουμε και στα πανεπιστήμια άλλωστε ως φαινόμενο, δηλαδή μπορεί να είναι πιο πολλές οι φοιτήτριε από ότι οι φοιτητέ στα πανεπιστήμια, ωστόσο καθηγητές είναι σε συντριπτικές πλειονότητες άντρε. Και άλλο ένα πρόβλημα, όταν βλέπουμε να δουλεύουν σε έναν κλάδο κατά πλειονότητα γυναίκες, χαρακτηριστικό είναι ότι τα επίπεδα των αμοιβών είναι χαμηλότερα από ότι σε κάποιο άλλο κλάδο. Εδώ κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να πω ότι όταν βλέπουμε πολύ περιορισμένη παρουσία των γυναικών στα ΜΜΕ, όντως μπορεί να πρόκειται για διάκριση, οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι κάτι το θετικό, αλλά ίσως θα ήταν καλό να κοιτάξουμε πιο αναλυτικά τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Γιατί δεν είναι αυτόματος ο συσχετισμός ή το συμπέρασμα ότι όσο πιο πολλές είναι οι γυναίκες που εργάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα είναι και καλύτερο το περιεχόμενο. Αυτή είναι η παγίδα την οποία θέλω να καταδείξω υπογραμμίζοντας ότι Ε, μπορεί να υπάρχουν τομεί στου οποίου εργάζονται πολύ λίγε γυναίκε και να μην μπορούμε να αλλάξουμε κάτι και μόνο αν αρχίσουν να εργάζονται όλο και περισσότερε γυναίκε μπορούμε να δούμε με τον καιρό όμω κάποιε αλλαγέ ενδεχομένω. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει και το βλέπουμε ήδη σε μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και αναπτύσσεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τσεχία να αλλάξει η νοοτροπία αυτό που λέμε κουλτούρα στα ΜΜΕ, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τις κοινοβουλευτικές, τις ε, κοινωνικές αξίες. Και βέβαια πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι τα ΜΜΕ δουλεύουν μέσα ένα, σε ένα και συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό ε, περιβάλλον. Όσο λοιπόν δεν έχουμε γενικότερα ευαισθησία στην κοινωνία μας σε σχέση με, τις, με τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, με την ισότητα των δύο φύλων, δεν θα αλλάξει η κατάσταση στα ΜΜΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Δακόκοβα. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ντονατέλα Μαρτίνη, που είναι διευθύντρια της οργάνωσης Donain Quota. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μας ε, προσκαλέσατε εδώ στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Σήμερα λοιπόν... Σήμερα λοιπόν αρχόμαστε ε, και εμείς εδώ ως ακτιβίστριες, ε, φεμινίστριες. Ας επικεντρωθώ λίγο τώρα σε αυτά που έχω να σας πω, που είναι πολλά για τα 15 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου. Η οργάνωσή μας, η Donen Quota, γυναίκες της ποσοστώσης δηλαδή, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, που είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οργάνωση ε, στην οποία περιλαμβάνονται πολλές επιμέρους οργανώσεις. Και το 2013 με την ε, γαλλική αντίστοιχη οργάνωση Sien de Garde, δημιουργήσαμε την WICAMS, που είναι ένας συνασπισμό ευρωπαϊκών ομάδων που αγωνίζονται κατά του σεξισμού στα μέσα ενημέρωσης, στα πλαίσια δηλαδή και τη ε, σύμβαση του ΟΙΕ. Θέλουμε να αποφύγουμε τις διακρίσεις λοιπόν στα μέσα ενημέρωσης. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η νομοθεσία κατά του σεξισμού στα μέσα ενημέρωση. Και αυτό με την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκδοση μιας οδηγίας. Τι χρειαζόμαστε αυτή την οδηγία. Θα επικεντρωθώ στην περίπτωση της Ιταλίας. Γιατί δείχνει τι συμβαίνει και παντού στην Ευρώπη, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση τη Γαλλία. Γιατί η Γαλλία πρόσφατα υιοθέτησε πολλά μέτρα, κυρίως στον τομέα της διαφήμισης, κατά ε, του σεξισμού. Στις αρχές Ιουλίου λοιπόν η Επιτροπή ΣΥΤΑ και κυβερνητικά όργανα επίσης ασχολήθηκαν με τις διακρίσεις κατά των γυναικών. Ευχαρίστω να σας διαβάσω λοιπόν τι λέει η έκθεσή μας. Είμαστε μέσα σε ένα δίκτυο οργανώσεων της Ιταλίας για τα δικαιώματα των γυναικών, η οποία καταπολεμά τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στις διαφημίσεις. Σε αντίθεση με άλλε ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία δεν έχει νομοθεσία για να αντιμετωπίσει στερεοτυπικές συμπεριφορές και σεξιστικές από τα μέσα ενημέρωσης. Από το 2010 Προτάθηκαν διάφορα νομοσχέδια, αλλά χωρίς να προχωρήσει τίποτα. Από το 2011 και σε παραβίαση της σύμβασης του ΟΗΕ του άρθρο για την ε, καταπολέμηση των διακρίσεων, συστάσεις 24-25 κλπ, προκειμένου να συμπεριληφθεί το θέμα των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στην διαφήμιση, όπως ακριβώς λέει η σύμβαση, είχαμε ένα έκτακτο εθνικό σχέδιο δράσης κατά του σεξισμού και της βίας σε βάρος των γυναικών με την πρωτοβουλία της Τζοβάνα Μαρτέλη που δούλευε υπό τον Πρωθυπουργό Ρέντσι και πρότεινα να δημιουργηθούν πάνελς με εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα ελέγχουν τις επιπτώσεις των σεξιστικών συμπεριφορών που έχουν να κάνουν με την εκπροσώπηση των φίλων. Δεν υπήρξε όμως καμία ένδειξη όσον αφορά τα κριτήρια τα οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία τέτοιων πάνελ. Το σχέδιο πάντως δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Και αν συγκρίνουμε με τα όσα είχαμε στην Σιωδέξη του 2011, δεν υπάρχει καμία υπηρεσία ελέγχου από πλευράς της κυβέρνησης που ελέγχει τα στερότυπα αυτά και πώς αντικατοπτρίζονται οι γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης γενικότερα και την ε, διαφήμιση ειδικότερα. Υπάρχουν ε, τρεις υπηρεσίες ελέγχου από την οργάνωση την Εθνική Δημοσιογράφων, την Ατζικόμο που είναι μια υπηρεσία που ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης και από την ΡΑΙ, την ε, κρατική τηλεόραση. Οι δύο πρώτες περιπτώσεις δεν δημοσιοποιούν τα συμπεράσματά τους, ενώ η ΡΑΙ το κάνει χωρίς όμως να προβλέπει διορθωτικά μέτρα ή κυρώσεις. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το CSA πριν από μερικές ε, μέρες σε σχέση με την ε, ΔΕΟΤ ε, κατηγορήθηκε για προγράμματα τέτοια σεξιστικά. Μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα λοιπόν ότι δεν υπάρχει νομικό ή άλλο κατάλληλο μέτρο που να έχει οθετηθεί μέχρι σήμερα για να διασφαλίσουμε ότι τα δημόσια ε, δίκτυα, τα ραδιοτηλεοπτικά φροντίζουν να τηρούν με τα μέτρα αυτά την σύμβαση του ΟΗΕ. Δεν συμβαίνει καθόλου κάτι τέτοιο. Αντίθετα υπάρχουν πρακτικές που οδηγούν σε διακρίσεις σε βάρος των ε, γυναικών συστάσει. Τώρα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό ορισμό του ότι είναι σεξιστική διαφήμιση. Δεύτερον, πρέπει να ευθετηθεί νομοθεσία που να καταπολεμά τα στερεότυπα και τι σεξιστικές συμπεριφορέ στα μέσα ενημέρωση και την διαφήμιση. Και τρίτον, πρέπει να υπάρξει ένας ανεξάρτητος μηχανισμός ad hoc με αποτελεσματική βέβαια πρικοδότηση και επάνδρωση και με κατάλληλες κυρώσεις που να προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις. Η αναποτελεσματικότητα του μηχανισμού αυτορύθμισης όσον αφορά τις αξιστικές συμπεριφορές στα μέσα ενημέρωσης και την διαφήμιση είναι κάτι που μας κάνει να λέμε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Όπως αναφέρει και η κυβερνητική έκθεση, η μόνη δυνατότητα δράσης κατά σεξιστικής διαφήμισης είναι να αναφέρεται κανείς σε, στον φορέα που ονομάζεται IAP και που είναι ε, η υπηρεσία αυτορύθμισης όσον αφορά την ε, διαφήμιση. Κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί ότι δεν φτάνει για την καταπολέμηση των σεξιστικών ε, διαφημίσεων. Έτσι κι αλλιώ δεν έχει περάσει τελικά καμία νομοθεσία όπως είπαμε από το 2011, αλλά ακόμη και αν είχε συμβεί αυτό δεν θα ήταν αποτελεσματικό αυτό το μέτρο. Επίσης, Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την ε, ΟΥΠΑ που είναι οι χρήστες της διαφήμισης. Από το 2011 πάντως η ΑΚ δεν περιλαμβάνει ειδικού για θέματα φύλου. Πώς λοιπόν θα καταπολεμήσουμε τις εξιστικές διαφημίσεις. Οι οργανώσεις των γυναικών προωθούν λοιπόν τα συμφέροντά του και τις επιθυμίες τους στους φορείς αυτούς και η μπορεί να δώσει συμβουλευτικά γνωμοδότηση χωρίς όμως να έχει καμία δυνατότητα να επιβάλλει τα συμπεράσματά της ή να επιβάλλει κυρώσεις για να σταματήσει κάποια σεξιστική διαφήμιση. Αν η εταιρεία που διαφημίζεται δεν θέλει να συμμορφωθεί, απλώ δεν συμμορφώνεται. Επίση, δεν έχει υπάρξει αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα της ε, συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι δήμοι της Ιταλίας μετά τη μελέτη του 2011 για να ελέγχεται η τοπική διαφήμιση. Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς εμφανίζονται οι γυναίκες ε, στους δημόσιου ραδιοτηλεοπτικούς ε, σταθμούς σας είπα, πρόκειται για τη ΡΑΗ. Σύμφωνα με την κυβερνητική έκθεση ΡΑΗ έχει οθετήσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για να βελτιωθεί η εικόνα της γυναίκας. Όμως, πρόκειται στην πραγματικότητα για κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά διάφορα φανταστικά σύριαλ που δεν μιλάει καν για το πώς πρέπει να αντικατοπτρίζεται η γυναίκα σε αυτές. Βλέπουμε λοιπόν αποτυχία εφαρμογής των γενικών κατευθυντήριων γραμμών, χωρίς όμως επιπτώσεις. Ούτε κυρώσεις, ούτε τίποτα άλλο. Το 2016 εξέπνευσε οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές της ΡΟΗ. Και στη συνέχεια ξεκίνησε μια διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών για να επιλεχθούν ποιες οργανώσεις θα συμμετέχουν σε ένα νέο σώμα αξιολόγησης. Δεν αναφέρεται τίποτα για πραγματογνωμοσύνη σε θέματα διακρίσεων. Παρά τις διαμαρτυρίες των οργανώσεων γυναικών. Πρόκειται για παραβίαση της σύμβασης και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να περάσουν πολλές διακρίσεις παρά τις αρχές που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση για 10 χρόνια. Σύμφωνα με τις παραχωρήσεις κάθε 5 χρόνια, στο παρελθόν κάθε 3 χρόνια, υπήρχε μια υπηρεσία για να ελέγχει την κατάσταση. Για την ανανέωση από το 2010 μέχρι το 2012, που ισχύει ακόμα, το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης απέτυχε να φροντίσει να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών στις διαβουλεύσεις. Και μόνο επειδή επέμειναν μη κυβερνητικές οργανώσεις των γυναικών, τελικά μπόρεσαν να συμπεριληφθούν σαν συνομιλητές εξού και εισήχθησαν 13 τροπολογίες. Τώρα για την επόμενη περίοδο, 2013-2015, οι, οι οργανώσεις των γυναικών πρότειναν πάλι τροπολογίες, οι οποίες εγκρίθηκαν ώστε κάθε σύμβαση να τηρεί τους όρους της σύμβασης. Ακόμα όμως κι αν προβλέπεται στην νομοθεσία δεν εφαρμόζεται και δεν υπάρχει μηχανισμός ο οποίος να φροντίσει οι τροπολογίες αυτές να περάσουν αυτόματα και στην επόμενη σύμβαση. Είναι θέμα βέβαια πολιτικής ε, βούλησης του Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης. Η απουσία κατευθυντήρων γραμμών λοιπόν όσον αφορά την εικόνα της γυναίκας είναι κάτι το οποίο έχει πιστοποιηθεί. Παρόλο που θα έπρεπε, γιατί προβλέπεται και στον προπολογισμό, η αρχή για τον τομέα, η Ατζικόμ, κάνει κάποιους ελέγχους όσον αφορά τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, αλλά χωρίς να δημοσιοποιεί τα απορίσματα και ούτε τα χρησιμοποιεί για δράσεις προς βελτίωση. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με τις προηγούμενες εκθέσεις γιατί τόσο η κυβέρνηση Μόντι όσο και οι επόμενες ακύρωσαν τα πάνελ εμπειρογνωμόνων που υπήρχαν από το 2012 στο τμήμα ίσων ευκαιριών προκειμένου να εκπονηθεί ένας κώδικας αυτορύθμισης με κατευθυντήριες γραμμές για την εικόνα των γενικών στα μέσα ενημέρωσης. Συστάσεις. Πλήρης εφαρμογή του CEDAW. Να εγκριθεί μια στρατηγική που θα εξετάζει τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης για το κατά πόσο ε, έχουν στερεότυπα σε βάρος των γυναικών. Να δημιουργηθεί επίσης ένας κώδικας διοντολογίας για σεξιστική εικόνα των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Επίσης, να υπάρξει απαγόρευση για οποιαδήποτε διαφήμιση που ελοχεύει διακρίση σε βάρος των γυναικών. Επίσης, να υπάρξει υποχρεωτικά η εισαγωγή ρητρών για τα δύο φύλλα στις δημόσιες ε, συμβάσεις της ΡΑΗ για παράδειγμα και αυτό να γίνει σε συνεργασία με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και μη κυβερνητικές οργανώσεις των γυναικών και να προσφέρουμε ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο για να παρακολουθεί τις ίσες ευκαιρίες ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών με τη συμμετοχή οργανώσεων γυναικών και του ΝΤΙΟ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σόντροβα για... που συμπεριέλαβε ένα άρθρο το οποίο έστειλα στη γραμματεία. Γιατί το λέω αυτό επειδή τον έφερε στο βιντεοσκοπημένο της μήνυμα. Πρόκειται για την ελευθερία έκφρασης όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων και το έχει γράψει η Εύα Μαρία Σβένσον, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της ε, Νορβηγίας και η Μαρία του Πανεπιστήμιου του Γκέτεμπουργκ. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζοντας ε, το άρθρο αυτό, βλέπει κανείς ότι μπορεί να συμφωνήσει μαζί μας για το ότι η ελευθερία έκφρασης, πώς να το πω, δεν πλήττει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αν δεν το αντιληφθεί κανείς σαν λογοκρισία. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Δονατέλα Μαρτίνη για την παρουσία σας, παρουσίασή σας, τις συστάσεις και τις προτάσεις σας. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην τρίτη καλεσμένη μας, τη Μαρτίν Σιμονής, που είναι Γενικός Γραμματέας, Γενική Γραμματέας της Βελγικής Ένωσης Επαγγελματιών Δημοσιογράφων. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι νομικός και γενική γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης ε, ε, Δημοσιογράφων του Βελγίου που ασχολείται με θέματα φύλων και ισότητας ε, στις ειδήσει. Δεν σας μίλησω για διαφημίσεις ή προγράμματα αναψυχής, αλλά για την παρουσία και τη θέση της γυναίκας στην ιδιοσιογραφία και πώς προβάλλονται οι γυναίκες στις ειδήσει. Έχω χωρίσει την ε, ομιλία μου σε δύο τμήματα. Το πρώτο θα το δούμε εντάχει, αφορά την παρουσία και την ε, προβολή, η παρουσίαση των γυναικών στα ΜΜΕ και κυρίως ε, στα δελτία ειδήσεων. Όταν ανοίγουμε τηλεόραση και βλέπουμε ειδήσει, πού είναι οι γυναίκες, πώς παρουσιάζονται. Έχουμε σχετικά πρόσφατες μελέτες πέραν του Global Media Monitoring Project που αναφέρθηκε προηγουμένω, που επίση είναι σημαντικέ για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Παρακολούθηση των ΜΜΕ, και δυστυχώ καταλήγουμε σε, στις ίδιες διαπιστώσεις. Θα κάνουμε λοιπόν μια παρουσίαση αυτών των διαπιστώσεων και θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα στις δράσεις. Γιατί μερικές διαπιστώσεις ε, ε, δεν είναι και πολύ ικανοποιητικέ. Επίση, θα δω πώ ε, συντίθενται τα, οι δημοσιογραφικέ ομάδε, ποια είναι η σύνθεσή του, πόσε γυναίκε συμμετέχουν σε τέτοιε δημοσιογραφικέ ε, ομάδε. Και θα αναφερθώ και στην βία στο χώρο εργασία και στην παρενόχληση στον κυβερνοχώρο μέσω του διαδικτύου των γυναικών δημοσιογράφων. Πού βρίσκονται οι γυναίκες λοιπόν στις ειδήσει στα δελτία ειδήσεων. Ναι. Έχετε εδώ δύο πίνακες. Ο πρώτος δείχνει τη θέση των γυναικών ε, στο ημερήσιο τύπο και βλέπετε μόλις 17%. Όταν ανοίγετε την εφημερίδα σας δηλαδή, αυτό ε, προβλέπει μια βελγική έρευνα για, για γαλλόφωνες εφημερίδες, βλέπουμε μόνο 17%. Δεν μιλούμε για γυναίκες δημοσιογράφους, για τη φωνή των γυναικών στις ειδήσει, στις, ε, στις εφημερίδες, μόνο 17%. Στην τηλεόραση είναι κάπως καλύτερη θέση των γυναικών, φτάνουμε στο 37% με βάση τις μελέτες, άλλοτε μιλούμε για 30% και άλλοτε για 40%. Αυτά ως προς τα δελτία ειδήσεων. Τώρα για τα προγράμματα αναψυχής, εκεί είναι πιο εμφανής η παρουσία των γυναικών. Και μάλιστα σας έχω βάσει, ε, βάλει εδώ και το link, γιατί είναι και διαθέσιμε στο διαδίκτυο σχετικές μελέτες. Αν εξετάσουμε τώρα το ρόλο των γυναικών στα δελτία ειδήσεων, στην ενημέρωση, Βλέπετε στην πρώτη γραμμή ε, τις ε, κομπάρσους και τους κομπάρσους. Βλέπουμε ότι ε, καθημερινά και στον τύπο και στα δελτία ειδήσεων ή στην ενημέρωση οι περισσότερες γυναίκες είναι κομπάρσοι και κυρίως σε ομάδες. Δεν φαίνονται καν συγκεκριμένα. Και στη δεύτερη γραμμή έχουμε τη, την εμπειρογνωμοσύνη. Έχουμε πολύ συχνά στα ΜΜΕ συνεντεύξει με εμπειρογνώμονε. Όταν όμω έχουμε τέτοιες συνεντεύξει, ποιοι είναι οι περισσότεροι εμπειρογνώμονε, Έγινε μια ε, καταμέτρηση των εμπειρογνωμόνων και βλέπουμε ότι στα καθημερινά ΜΜΕ 9 ε, στους 10 εμπειρογνώμονες που δίνουν συνέντευξη είναι γυναίκες, δηλαδή ε, άντρες, συγγνώμη. 96% των εμπειρογνωμόνων που καλούνται να δώσουν συνέντευξη είναι άντρες. Τώρα, βλέπουμε την κατανομή των ανδρών και των γυναικών ανάλογα με, το, με την ηλικία τους. Όταν θέλουμε να προσδώσουμε μια ηλικία σε κάποιον που βλέπουμε στο, στα μίδια, στα ΜΜΕ, βλέποντα τη φωτογραφία του για παράδειγμα σε ένα άρθρο, τι παρατηρούμε ότι αν οι γυναίκε δεν είναι γύρω στα 20, γιατί έχουμε κυρίω παιδιά και έφηβες, και μέχρι τα 20 έχουμε μια ισότητα στην παρουσίαση ανδρών και γυναικών. Μετά που αφού παίρναν την ηλικία των 20, όταν γίνονται δραστήριε δηλαδή γυναίκε, εξαφανίζονται από την ενημέρωση οι γυναίκε. Ενώ οι ενεργοί άντρε καταλαμβάνουν ε, το χώρο τη ενημέρωση. Επίση, οι ηλικιωμένε γυναίκε, όπω είπε και η προλαλήσασα, ε, οι ηλικιωμένε γυναίκε αυτέ εξαφανίζονται πλήρω από την ενημέρωση. Παρόλο που οι ηλικιωμένε γυναίκε είναι πολύ περισσότερε από του ηλικιωμένου άντρε, γιατί εκεί έχουμε αντιστροφή τη ηλικιακή πυραμίδα. Οπότε θα έπρεπε να, να ανατρέψουμε την κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών για να έχουμε μια ισορροπημένη αντανάκλαση και εκπροσώπηση της κοινωνίας. Τώρα βλέπουμε πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες στα διάφορα θέματα της ενημέρωσης. Στην τρίτη γραμμή βλέπετε τον αθλητισμό. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στον αθλητισμό που θεωρείται και αυτό το τμήμα της ενημέρωσης είναι θέαμα αλλά είναι και ενημέρωση. Βλέπετε ότι στον αθλητισμό 6 με 7% μόνο η παρουσία των γυναικών. Μόνο. Δηλαδή είναι η κατηγορία της ενημέρωσης ε, που πραγματικά κρατάει αφανή στις γυναίκες μαζί με την πολιτική και οικονομική δυσιογραφία. Ο αθλητισμός ε, έχει πολύ χαμηλή παρουσία των γυναικών. Επίσης, κατανομή των φύλων με βάση τον προσδιορισμό τους. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια, αν θέλετε. Διερωτηθήκαμε λοιπόν, είναι ίσοι άνδρες και γυναίκες ε, στην ε, αναγνώρισή τους, ε, στον προσδιορισμό τους, ε, με ονοματεπώνυμο, με επάγγελμα. Όταν βλέπουμε την κατηγορία των ανθρώπων που δίνουν συνέντευξη και όταν προσδιορίζονται μόνο από το μικρό του όνομα, οι είναι, οι περισσότερες είναι γυναίκες. Όταν έχουμε κατηγορία που αναγνωρίζεται με βάση το ονοματεπώνυμο και το επάγγελμα, τότε η συντριπτική πλειοψηφία είναι άντρες. Οπότε δεν είναι ίσοι άντρες και γυναίκες ε, στο, στην αναγνώρισή τους και στον προσδιορισμό τους. Όταν το επισημαίνουμε στους δημοσιογράφους μας λένε όχι αποκλείεται, εμείς δεν δουλεύουμε έτσι. Κι όμως οι μελέτες αυτό αποδεικνύουν. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιου είδους μελέτες. Γιατί αισθηκτοδός πραγματικά ε, δεν θα βλέπαμε διαφορά στην αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών από τους δημοσιογράφους. Και όμως αυτό δείχνουν οι μελέτες, ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Οι άντρες παρουσιάζονται πιο επώνυμα. Επίσης, ε, δυστυχώς ε, συγκλίνουν οι διαπιστώσεις ε, των αριθμών μελετών που δείχνουν ότι ελάχιστα εκπροσωπούνται οι γυναίκες στην ενημέρωση. Είναι αφανής κυρίως στην αθλητική πολιτική και οικονομική ειδησιογραφία, όπως σας είπα. Έχουν κυρίως ρόλους κομπάρσου. 9 στους 10 εμπειρογνώμονες που δίνουν συνεντεύξεις, επαναλαμβάνω, είναι άντρες. Και επίση ε, δεν αναγνωρίζονται, δεν προσδιορίζονται επώνυμα οι γυναίκε ε, ούτε ισότιμα παρουσιάζονται στην ενημέρωση. Αυτό γίνεται μόνο μέχρι τα 20 του. το ότι υπάρχει ίση εκπροσώπηση. Μετά εξαφανίζονται. Αυτέ λοιπόν είναι οι συχνέ διαπιστώσει των μελετών. Ε, και λέμε γιατί να αλλάξουν τα πράγματα, μα πρέπει να αλλάξουν γιατί τα μίντια μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της νοοτροπίας. Και θα πρέπει να αλλάξουμε τη σκοπιά μας, να επικεντρωθούμε στην ποιότητα της ενημέρωσης γιατί είναι απαράδεκτο να μιλάνε τόσο λίγο ή τόσο άσχημα για το μισό του πληθυσμού οι δημοσιογράφοι. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στις διαπιστώσεις, θα πρέπει να περάσουμε στη δράση. Και θα σας παρουσιάσω εδώ κάποιες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει. Πριν περάσω όμως στις πρωτοβουλίες, θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε και να κάνω κάποιες συστάσεις ή προτάσεις, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις μελέτες, τεκμηριωμένες μελέτες περιεχομένου, γιατί συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών. Όταν δείχνουμε στον κόσμο πώς διαμορφώνεται η πληροφορία, μερικές φορές ε, υποσυνείδητα, τότε ε, ο κόσμος συνειδητοποιεί καλύτερα το πώς δουλεύει η δημοσιογράφη και ίσως έτσι δημιουργηθεί η ανάγκη της αλλαγής. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις φοιτήτριες δημοσιογραφίας και να τις ευαισθητοποιήσουμε για αυτά τα θέματα, γιατί ε, δύο τρίτα των, των φοιτητών δημοσιογράφων είναι κορίτσια. Αυτές θα πρέπει πρώτα να προσεγγίσουμε. Επίσης, να συνεργαστούμε με δημοσιογράφους και διευθύνσεις ΜΜΕ μέσω των ε, μόνιμων ε, ομάδων και επίσης να κάνουμε ποσοτικοποιημένες αναλύσεις, δηλαδή κάθε μέσο μαζικής ενημέρωση να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Κάτι που είναι δύσκολο οικονομικά αν υπάρχουν ε, κάποια εσωτερικά ευρωβαρόμετρα από τις υπηρεσίες ε, και οργανισμούς οπτικοακουστικών μέσων. Θα πρέπει τέτοιες πρωτοβουλίες να τις εθαρρύνουμε και να τις επεκτείνουμε, ώστε ενδεχομένω να εκπονήσουμε και κάποια σχέδια ε, ισότητας με ποσοτικοποιημένους δείκτες και σχέδια δράσης. Θα σας παρουσιάσω τώρα το μηχανισμό που αναπτύξαμε για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους στο Βέλγιο. Πρόκειται για το, μια βάση δεδομένων που λέγεται Εξπερτάλια. Είναι βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων ε, διαφορετικής προέλευσης. Εδώ δίνουμε έμφαση στην πολυμορφία και στη διαφορετικότητα. Άνδρες και γυναίκες διαφορετικής προέλευσης. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων που επιτρέπει στους δημοσιογράφους να έχουν ένα εργαλείο στα χέρια τους για να μην έχουν την δικαιολογία και να λένε ότι θέλουμε πολύ ευχαρίστως να καλέσουμε σε συνέντευξη γυναίκες εμπειρογνώμονες, αλλά τι βρίσκουμε. Ε, ορίστε, έχετε τη βάση δεδομένων για να τι βρείτε. Πολύ χρήσιμο λοιπόν εργαλείο και για του δημοσιογράφου αυτή η βάση δεδομένων. Και επίση ανταποκρίνεται με ρεαλιστικό τρόπο σε αυτή την δικαιολογία που μα φέρουν οι δημοσιογράφοι ότι δεν βρίσκουν γυναίκε εμπειρογνώμονες. Εδώ του αποδεικνύουμε ότι υπάρχουν και του επιτρέπουμε να κάνουν μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση των δημοσιογραφικών του πηγών και να δώσουν έμφαση στην διαφορετικότητα και στην πολυμορφία των πηγών και της προέλευσης. Αν κάνουμε μια έρευνα σε αυτή τη βάση των δεδομένων με μια λέξη κλειδί φύλλο, θα μπορούσα να είχα βάλει άλλη λέξη, μαθηματικά ή αρχιτεκτονική, βλέπουμε αμέσως να ε, εμφανίζονται 12 γυναίκες εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί, οπότε οι δημοσιογράφοι έχουν πρόσβαση στα βιογραφικά τους και επίσης και στα προσωπικά τους στοιχεία εφόσον εγγραφούν. Και μάλιστα κάνουμε ένα coaching για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα είδος προπόνησης και καθοδήγησης για, τις, για τους εμπειρογνώμονες, για να τους ε, εκπαιδεύσουμε να μιλούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να γίνουν καλές, καλοί πελάτες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού θα ξέρουν να απευθύνονται στο κοινό, θα ξέρουν να μιλάνε. Να λοιπόν, τους βοηθούμε να αναπτύξουν τέτοιες δεξιότητες. Τέτοια τους εργαλεία είναι εύκολο να αναπτυχθούν. Επίσης, ε, υπάρχει και νομοποίηση γιατί εκπηγάζουν από την ίδια την Ένωση των Δημοσιογράφων. Δεν είναι μια εξωτερική οργάνωση που υποδεικνύει στους δημοσιογράφους πώς πρέπει να εργαστούν. Ο ίδιος ο κλάδος, το ίδιο το επάγγελμα, το ίδιο το ε, σωματείο τους επιλήφθηκε του θέματος. Επίσης, ε, για την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου στηριχθήκαμε σε μελέτες περιεχομένου, οπότε είναι ηρθολογική μελέτη. Δεν ξεκινήσαμε με κάποιες ε, ε, αισθηκτόδης απλώς σκέψης και στόχος του εργαλείου είναι να αποφύγουμε και τις αξιολογικές κρίσεις γιατί θα πρέπει να αποφύγουμε να ε, πούμε στους δημοσιογράφους δεν δουλεύετε σωστά, εμείς θα σας δείξουμε πώς θα το κάνετε. Απλώς να τους παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, να τους ρωτήσουμε τι είναι κατά τη γνώμη μας σας ποιοτική ενημέρωση και πώς θα καταλήξουμε σε τέτοια ποιοτική ενημέρωση. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σωστό εγχείρημα που χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό στόχος πολύ σημαντικός, αν θέλουμε πραγματικά να προωθήσουμε αυτό το θέμα, να κάνουμε τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους συμμάχους ε, στον αγώνα μας για την ισότητα των δύο φύλων και την ισοτιμία. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κέριο ρόλο γιατί είναι ένα σκαθρέφτης της εικόνας της κοινωνίας αλλά δημιουργούν και νέες εικόνες ενίσχυσης ε, και καταπολέμηση των στερεοτύπων ανάλογα με τη θέση που θα λάβουν. Και φτάνουμε εδώ στο δεύτερο τμήμα της ομιλίας μου για να σας δείξω πού βρίσκονται οι γυναίκες στις, ε, στη σύνταξη. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από μια βελγική μελέτη που έγινε το 2013 και αφορά όλη τη βελγική επικράτεια και έχουμε στο ανοιχτό γαλάζιο τις γυναίκες, ε, στο σκούρο γαλάζιο τους άντρες και με ηλικιακή κατανομή και βλέπετε πως η κατανομή δεν είναι ισότιμη ανάλογα με το, την ηλικία του στα διάφορα επαγγέλματα. Και βλέπουμε ότι ε, στα 35 από αφιπηρετούνται κατά κανόνα οι γυναίκες, που είναι μια επιλογή τους, ε, γιατί εκεί, σε εκείνη την ηλικία, στα 35, καλούνται να κάνουν μια επιλογή. Θα παντρευτούν, θα κάνουν παιδιά, θα βρουν σύντροφο. Και πραγματικά η δημοσιογραφία είναι ένα χρονοβόρο επάγγελμα και απορροφά όλο το χρόνο και τη ζωή του δημοσιογράφου. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει μία απάντηση στο πώς θα συνδυάσει όλες αυτές τις επαγγελματικές ή τις προσωπικές υποχρεώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, την εκπροσώπηση των γυναικών στην ιεραρχία, στις υψηλόβαθμες θέσεις. Αν δούμε τους μάνατζερ, βλέπουμε ότι έχουμε τριπλάσιο, τετραπλάσιο αριθμό ε, διοικητικών ανώτατων στελεχών ε, σε άντρες. Ε, και στις ε, Διάμεσέ διοικητικέ θέσει πάλι οι άντρε είναι πολύ περισσότεροι. Σε ό,τι αφορά τη σταδιοδρομία, βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο 15 χρόνια σταδιοδρομία, ενώ οι άντρε 19. Επίσης, βλέπουμε ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι ε, Συνήθω έχουν, δεν έχουν παιδιά σε σχέση με τους άντρες. Οι πολύ λιγότερε γυναίκες δημοσιογράφοι έχουν παιδιά από ότι οι άντρες συναδελφοί του. Επαναλαμβάνω, αυτό το επάγγελμα απαιτεί πλήρη αφοσίωση, είναι τελείως χρονοβόρο και απαιτεί κάποιε ε, επιλογές ζωής. Και οι εργασιακές συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες και πολύ συχνά εμποδίζουν και σίγουρα εμποδίζουν για τις γυναίκες τη συνύπαρξη της προσωπικής και της επαγγελματική ζωής. Και αυτό, αυτή η αδυναμία συμφιλίωσης αγγίζει περισσότερο τις γυναίκες. Και αν μου επιτρέπετε και πάλι να κάνω κάποιες συστάσεις, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή και επιστημονική διάγνωση των εμποδίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία, κάθε είδου ε, προβλήματα και εμπόδια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη που συνδέονται με τι εργασιακέ συνθήκε και το δημοσιογραφικό περιβάλλον και με βάση τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εκπονήσουμε ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράση με ποσοτικοποιημένου δείκτε για να δούμε κατά πόσο βελτιώνονται τα πράγματα. Επίση, να ευαισθητοποιήσουμε τι φοιτήτριε και τι νέε γυναίκε δημοσιογράφου για τι ανισότητε που θα αντιμετωπίσουν στο χώρο εργασία και κυρίω στι μισθολογικέ διαφορέ και να προτείνουμε κατάλληλε αντιδράσει και λύσει μέσω των διαπραγματεύσεων. Επίσης να στηρίξουμε τις δράσεις ε, καθοδήγησης ε, ή ορισμού μέντορα. Υπάρχουν ε, ενδιαφέρουσε πρωτοβουλίες στη Γερμανία στο δημοσιογραφικό κλάδο, επίσης πρωτοβουλίες μόνιμης κατάρτισης, διαβίου κατάρτισης και να αναλύσουμε και τα νέα ζητήματα που θέτει η ψηφιοποίηση και κυρίως η παρενόχληση των γυναικών δημοσιογράφων στο διαδίκτυο. Έχουμε εδώ μία εκστρατεία στην ε, Ασία κατά της ε, παρενόχλησης στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο. Μπορείτε να διαβάσετε αυτή την, ε, να δείτε τα στοιχεία αυτής της εκστρατείας για τα ανησυχητικά ποσοστά, πολύ εντυπωσιακά και ανατοχιαστικά ποσοστά εμφάνισης της παρενόχλησης στο διαδίκτυο κατά των γυναικών κυρίως δημοσιογράφων. Επίσης θα πρέπει να επενδύσουμε στην κατάρτιση και επιμόρφωση των επαγγελματιών και των φοιτητών και να ευαισθητοποιήσουμε για τα όργανα αυτορύθμισης, τα Συμβούλια Διοντολογίας. Πριν από λίγο το αναφέραμε για την διαφήμιση. Εγώ το διαπιστώνω και στην ενημέρωση. Θεωρώ ότι ακόμη τα Συμβούλια Αυτορύθμισης δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί δεόντως για θέματα σεξισμού. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με αυτά τα όργανα αυτορύθμισης για τα θέματα αυτά. Δεν έχουμε πρόσφατες ποσοτικοποιημένες μελέτες για τη μισθολογική διαφορά στις εφημερίδες, στα ΜΜΕ, ούτε πρόσφατες μελέτες για την παρουσία των γυναικών στη σύνταξη των ΜΜΕ. Να σας δείξω όμως μια νέα εκστρατεία που γίνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και αφορά τη βία στο χώρο εργασίας στα γραφεία σύνταξης δηλαδή ουσιαστικά. Φυσικά δεν θα πρέπει να γενικεύουμε, αλλά τα στοιχεία που μας δίνει αυτή η μελέτη για την σεξιστική βία στο χώρο εργασία, δυστυχώ αυτά τα στοιχεία είναι πολύ εντυπωσιακά. Ένα τέταρτο των γυναικών που απασχολούνται στα μέσα μαζική ενημέρωση έχουν υποστεί σωματική βία στο χώρο εργασία ή στο εγγύς περιβάλλον. Οι μισέ γυναίκε που απασχολούνται στα μέσα μαζική ενημέρωση έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και τρία τέταρτα των γυναικών που δουλεύουν στα ΜΜΕ έχουν υποστεί εκφοβισμό, απειλέ ή και κακή μεταχείριση. Δυστυχώς δεν ε, έχουμε επίγνωση ή συνείδηση της έκθεσης αυτού του φαινομένου και αυτής της πραγματικότητας. Σας έδωσα τα στοιχεία ε, στο PowerPoint της εκστρατείας αυτής. Θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Θέλουμε μία Διεθνή Σύμβαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας για την καταπολέμηση της εξιστικής βίας στο χώρο εργασίας. Και έρχομαι εδώ σιγά σιγά προς το τέλος της ε, ομιλίες μου και να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή. Σας ευχαριστούμε κυρία Μαρτίν Σιμονής για την παρουσίαση. Περνάμε στη συζήτηση. Έχετε το λόγο για ερωτήσεις, σχόλια και το καθεξής. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χάνεμπολ, για τις πολύ λεπτομερείς αυτές ε, παρουσιάσεις. Όντως, είναι πολύ απογοητευτικό το να βλέπουμε πόσος δρόμος μας μένει ακόμη και μάλλον τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν είναι, δεν είναι αυτά που παρουσιάζουν τη χειρότερη κατάσταση γενικά. Βλέπουμε τις συνθήκες αυτές τη βάρος των γυναικών σε όλου του τομεί απασχόληση, όπω άλλωστε ξέρουμε εμεί εδώ πολύ καλά. Ε, αναφερθήκατε σε συγκεκριμένου φραγμούς όμω ε, στην ε, ε, παρουσία των γυναικών στα ΜΜΕ. Πολλά βέβαια θα είναι τα προβλήματα σχετικά με το συνδυασμό του επικοινωνικού με τον, οικογενειακό βίο, όπως ότι οι δημοσιογράφοι συχνά θα έχουν ε, δυσκολίες ε, γιατί ένας ρεπόρτερ Φερπίν πρέπει να ταξιδεύει σε μακρινές περιοχές, δεν μπορεί να αφήνει την οικογένειά του. Ε, τα βλέπουμε και εμείς αυτά εδώ πέρα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας παρουσιάσατε και Χαίρομαι που τουλάχιστον συζητιούνται τα θέματα του συγκερασμού του επαγγελματικού με τον οικονομικό βίο. Και σε σχέση με την ηλικία, όντως βλέπουμε σε διάφορα επαγγέλματα ότι έρχεται μια ηλικία όπου μειώνεται ε, η παρουσία των γυναικών στον ε, επαγγελματικό χώρο. Και γι' αυτό θα ήταν καλό να κοιτάξουμε ιδιαίτερα τα θέματα της ε, φροντίδας για τα παιδιά κτλ. Για να μπορούν οι γυναίκες να εργάζονται και όταν έχουν οικογένεια και παιδιά. Ωστόσο υπάρχει και το θέμα των πιο ηλικιωμένων γυναικών με ιδιαίτερα οξυμένη μορφή στα ΜΜΕ, αλλά όχι μόνο στα ΜΜΕ Και το επάγγελμα του δημοσιογράφου έχει να κάνει με το τι δείχνουμε στον κόσμο. Και άρα βεβαίως έχει σημασία η εμφάνιση γενικά για τις γυναίκες, αλλά και ιδιαίτερα στο χώρο της δημοσιογραφίας. Γιατί η εμφάνιση μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τον τρόπο που σκέφτονται οι θεατές στο κοινό. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η διάσταση της εμφάνισης και για τους πολιτικούς τώρα με βεβαίως αυτό. Και πρέπει να το κοιτάξουμε γιατί και από, και από, τα, από τα μέσα μάλλον κυρίως μαζικής ενημέρωσης ενημερώνονται ε, οι πολίτες για την οικονομία, για την κοινωνία κτλ. Πολύ περισσότερο μάλιστα από τα ΜΜΕ από ότι από τους πολιτικούς τους ίδιους. Επομένως μπορεί να μιλούμε για την παρουσία γυναικών στις ηγετικές πολιτικές θέσεις αλλά πρέπει να κοιτάξουμε οπωσδήποτε και αυτή τη διάσταση της δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ. Επίσης πρέπει να το κοιτάξουμε και σε αναλογία με τη σύνθεση του πληθυσμού. Εφόσον ο πληθυσμός και θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη αναλογία παρουσίας γυναικών πιο ηλικιωμένων στα ΜΜΕ. Ενώ βλέπουμε ότι συμβαίνει κάτι που ακολουθεί διαφορετικές τάσεις. Και έτσι στον Ηνωμένο Βασίλειο έγιναν κάποιες ε, εκστρατείες ευαισθητοποίησης στα θέματα των γυναικών και της ηλικία, χωρίς μεγάλη επιτυχία πρέπει να πούμε. Γιατί δεν μπορεί κανείς ε, και από τα ΜΜΕ να αγνοήσει τη διάσταση της ηλικία ε, των γυναικών δημοσιογράφων. Εν αυτό θα θέλω να μου πείτε, να μου εξηγήσετε λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ. Κύριος Μαχτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ τις ομιλήτριες, γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω ε, ολόκληρες τις ε, παρεμβάσεις. Οι δύο τελευταίες που παρακολούθησαν ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Η τελευταία δεν, τι μας δείχνει ότι ο καλλιεργημένος, ομορφωμένος κόσμος είναι εξίσου φαλοκρατικός και μισογενικός όπως κάθε άλλο τομέας της κοινωνίας. Εγκάρσιο λοιπόν το φαινόμενο και ακριβώς εδώ είναι που έρχεται ο κόμπος το χτένει και πρέπει να πούμε τι οφείλουμε να κάνουμε. Και βέβαια παραπέμπουμε πάντα σε ευθύνες των πολιτικών, στη συμπεριφορά, στην ορολογία που χρησιμοποιείται. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν υπάρχουν εφερειπίν ε, βουλευτές οι οποίοι απευθυνόμενοι στην προεδρεύουσα, όχι τη συγκεκριμένη πρόεδρο σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πρόεδρος γυναίκα σε μια επιτροπή και ακούμε να λένε κυρία πρόεδρος ή κυρία βουλευτή, βουλευτής, ε, Madame le Président ή Madame le Député, βάζουν δηλαδή το αρσενικό άρθρο στα γαλλικά. Ε, οπωσδήποτε υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Για να μιλήσω δε συγκεκριμένα για το χώρο της ε, τηλεόρασης, το παιδί μου που είναι τόσο μικρό μου είπε εδώ και χρόνια μάλιστα παρατήρησε ότι στα talk show πάντα κάθονται στις πρώτες σειρές όμορφες, νεαρές, χαμογελαστές νε, ε, κοπέλες με μεγάλο ντεκολτέ κατά προτίμηση. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν ο σεξισμός και ο μισογενισμός. Δεν βλέπω κανένα τηλεοπτικό συμβούλιο να αντιδρά ε, στο γεγονός ότι η γυναίκα καθίσταται προϊόν προς πώληση, προϊόν προώθησης ή κράχτης. Δυστυχώς πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτούς τους όρους. Και επίσης, ε, επειδή πρόσφατα και τις φιλευτικές εκλογές στη Γαλλία, γίνεται χαμός με το που βγήκε μια είδηση ότι έναν άντρα τον έδερνε η γυναίκα του. ε, συγγνώμη, ε, για, έναν άντρα υποψήφιο τον οποίον κέρδισε μια γυναίκα υποψήφια. Γιατί δεν βρήκε άλλο επιχείρημα ο κύριος αυτός παρά μόνο να πει τι αυτή που θα βγει βουλευτής τώρα πώς θα ασχοληθεί με τον άντρα της και τα παιδιά της. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν έχουμε μπορέσει να κάνουμε έναν, ε, ένα γομάρι το οποίο δεν διψάει να πάει στη βρύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε αυτή την ευαισθητοποίηση. Το δείξατε άλλωστε και με τα παραδείγματα που μας δώσατε από τα ΜΜΕ και, γενικά, και ειδικότερα τους δημοσιογράφους. Αλλά αυτό που είπατε να μετατρέψουμε σε συμμάχους μας τους δημοσιογράφους. Έστω θα το δεχθώ, αλλά με την εξής επιφύλη, με την φύλαξη. Δεν θα τους κάνουμε και ε, κολακία, δεν θα τους ε, γεμίζουμε με ε, φιλοφρονήσεις ή θα αγνοούμε τα λάθη που κάνουν γιατί αν χρησιμοποιούν μισογενικό ή φαλοκρατικό ε, σύστημα και διατυπώσεις δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό, θα τους πατάξουμε. Ε, για την έκθεση Λεκρή που είχαμε στην προηγούμενη ε, σύνοδο που μιλάει για τη διαφάνεια στα μισθού. ξέρετε ότι πλειοψηφία των βουλευτών τη δεξιά, αλλά όχι μόνο της δεξιάς καταψήφισε την έκθεση και η κυρία Λεγκρίπ ήτανε από την ε, δεξιά παράταξη. Και όμως οι συνάλφοι της παράταξής της την καταψήφισαν αυτή την ιδέα για, για πιο διαφανείς μισθούς. Με φαινόμενο λοιπόν ότι η μορφωμένη, καλλιεργημένη και τα λοιπά ανώτερη τάξη έχει εξίσου μισογενική κεφαλοκρατική στάση με οποιανδήποτε άλλη. Εγώ πιστεύω ότι πλέον πρέπει να εισαχθούν αυτοματοποιημένες κυρώσεις. Ξέρετε, εμένα μ' αρέσει να τρέχω γρήγορα με το αυτοκίνητο. Ε, και αυτό που με ανάγκασε να σταματήσω να πατάω τον γκάζι τόσο πολύ είναι το σύστημα με τους πόντους και με τα πρόστιμα πόντι στο δίπλωμα λοιπόν. Περισσότερο στη Γαλλία εφαρμόζονται παρά στο Βέλγιο τα συστήματα με τα ραντάρ που χρεώνουν στη συνέχεια έναν, δύο, τρει πόντους στο δίπλωμα και άμα, πει, άμα δει κανεί ότι κινδυνεύει να χάσει το δίπλωμά του τότε σταματάει να τρέχει και γρήγορα. Ε, λοιπόν, α είναι αυτοματοποιημένε οι κυρώσει ή σεξιστικέ ε, τοποθετήσει, παρατηρήσει κτλ. να καταστούν αδίκημα και άπαξ και ένα δίκημα να επιβάλλονται εξαιρετικέ κυρώσει. Τουλάχιστον για μένα αυτό πρέπει να συμβαίνει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Τώρα παρακαλώ τους ε, προσκεκλημένους μας, τις προσκεκλημένες μας να απαντήσουν. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να... Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αυτόματες απαντήσεις βέβαια δεν έχω. Να σας πω τι πρέπει να γίνει. Απλές λύσεις δεν υπάρχουν. Και έχω επισημάνει ήδη κάποιες ε, περιπλοκές και δυσκολίες σε σχέση με το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο ε, έντονη ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα ε, φύλλα στα ΜΜΕ. Στην Τσεχική Δημοκρατία, παραδείγματι, οι άντρες δημοσιογράφοι, δεν θα πω όλο και πιο συχνά βέβαια, αλλά ε, κι όμως είναι πιο πολύ σιγά σιγά οι άντρες δημοσιογράφοι οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα της ε, ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, προβάλλουν αυτό το μήνυμα εντός εισαγωγικών και όπως είπα δεν είναι μόνο γυναίκες αλλά και άνδρες δημοσιογράφοι και μάλιστα όχι μόνο δημοσιογράφοι αλλά γενικά και άνδρες σε θέσεις επιρροής. Επί παραδείγματι παραγωγή των ε, έργων, των ταινιών ενημέρωσης, ντοκιμαντέρ κτλ. Βλέπουμε να, επιβα... να πιέζουν προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, από την άλλη βέβαια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να τους αποθαρρύνουν από αυτήν την ε, προσπάθεια, προσπάθεια όπως είπα για δραστηριότητες σχετικές με την ισότιμη μεταχείριση. Χρειάζονται λοιπόν ε, πιο εντατικές δράσεις. Ας αρχίσουμε να μιλάμε περισσότερο για ε, όχι μόνο τον μέσο κοινό ε, πολίτη, αλλά και για όλους αυτούς που είναι ιδιαίτερες κατηγορίες. Είναι οι γυναίκες, είναι οι ανάπηροι, είναι τα άτομα ε, που ανήκουν στο χώρο ΛΟΑΔΜ και ούτω καθεξής. Αυτά όλα πρέπει να ανοίξουν και ας αντιληφθούν και οι άντρες ότι εάν δραστηριοποιηθούν στις δραστηριότητες και ρίξουν φως στα προβλήματα αυτά, μπορεί να κερδίσουν κιόλα σε απήχηση. Στην Τσεχία, εάν κάποιος ε, άντρας διαμαρτυρηθεί για το σεξισμό στις διαφημίσεις, παραδείγματι, του λένε «Μα δεν νιώθεις από αστεία». Γιατί θεωρείται ότι η παρουσίαση του γυμνού σώματος της γυναίκας μπορεί να είναι και χαριεντισμός. Άρα δεν έχει εσύ το χιούμορ αυτός που το βρίσκει κακό αυτό. Ε, πιστεύω πάντως για να ολοκληρώσω θα ήταν καλό οι άντρες που βρίσκονται σε θέσεις ηγετικές ε, να τοποθετηθούν ε, πρώτα απ' όλα. Παρακαλώ κύριε Μαρτίνη. Στην Ιταλία οι δημοσιογράφοι ακολουθούν, παρακολουθούν κάποια σεμινάρια κάθε χρόνο. Και κάθε φορά που παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα, τα σεμινάρια, έχουν κάποιο στόχο. Κάθε χρόνο δηλαδή πρέπει να πετύχουν κάποιο στόχο μετά από αυτά τα μαθήματα, αυτή την επιμόρφωση. Στην Ιταλία λοιπόν μπορεί να είναι εύκολο να υποχρεωθούν οι γυναίκες δημοσιογράφοι, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι ευαισθητοποιημένες όλες οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες να παρακολουθούν ένα μάθημα το χρόνο για θέματα ισότητας των δύο φύλων, κατά πολέμηση των διακρίσεων. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή δημοσιογράφους ευαισθητοποιημένους στο θέμα μετά από λίγα χρόνια. Όσον αφορά την ηλικία, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα επαγγέλματα στα μέσα ενημέρωσης και αλλού. Οι γυναίκες κάποια ηλικία δεν προβάλλονται πια. Είναι όπως και στην καθημερινή μας ζωή, στο δρόμο. Όταν είσαι νέα στην Ιταλία, τουλάχιστον, άμα είσαι νέα και όμορφη, έχεις πολλούς θαυμαστές στο δρόμο. Σε προσέχουν. Τώρα το λένε όχληση, αλλά όταν εγώ ήμουνα νέα δεν ήταν έτσι. Παρενόχληση το λένε σήμερα. Μετά τα 40 όμως πάει τελείως αυτό δεν, έχεις, δεν βλέπεις αυτή την εκτίμηση. Είναι κάτι πάντως πιο μεγάλο από αυτό που σκεφτόμαστε και ίσως θα έπρεπε να μελετήσουμε περισσότερο το τι συμβαίνει στην Ιταλία. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ τώρα εσείς, κυρία Μαρτίν Σιμονή. Ευχαριστώ. Θέλω να απαντήσω στην ε, ερώτησή σας γιατί εξαφανίζονται οι πιο μεγάλες ηλικία γυναίκες από τα δελτία ειδήσεων. Δεν έχω πολλές απαντήσεις ή προτάσεις, αλλά υπάρχει αυτό το φαινόμενο που θέλει νέες γυναίκες ε, στην τηλεόραση. Είναι κάτι που το παρακολουθούμε εδώ και καιρό. Βέβαια υπάρχει μια μικρή αλλαγή επειδή ακριβώς ε, οι γυναίκες που μπήκαν στη δημοσιογραφία πριν από χρόνια παραμένουν και μεγαλώνουν στην ηλικία. Πρέπει να μιλάμε και για τις καλές πρακτικές και υπάρχει μια σουηδική τηλεόραση, τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι το όνομά μπορώ να το βρω, που είναι περιφερειακή. Στόχος της ομάδας των δημοσιογράφων ήταν κάθε εβδομάδα να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα στους προσκεκλημένους τους. Έτσι λοιπόν σε ένα μήνα μέτρησαν και φρόντισαν να έχουν προσκαλέσει τόσους άντρες όσο και γυναίκες στις πολιτικές τους εκπομπές. Και πήγε καλά. Δεν υπάρχει υποχρεωτική ποσόστοση, δεν υπάρχει καμιά κύρωση από πίσω που να τους κυνηγάει, αλλά η διεύθυνση και οι ομάδες δημοσιογράφων αποφάσισαν να εφαρμόσουν αυτή την ισότητα στα πάνελ προσκεκλημένων. Και δούλεψε. Και αυτό ίσως θα λειτουργήσει καλύτερα, γιατί έχει επιπτώσεις και στο κοινό των θεατών. Είδαν ότι ανέβηκε η κροματικότητα πέντε μονάδες ε, στις γυναίκες. Και ακριβώ αυτό θα σώσει την παρουσία των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά το γεγονός ότι οι πιο μεγάλες στην ηλικία παρακολουθούν ε, τις ειδήσει, γενικά την τηλεόραση πολύ περισσότερο από τους νέους, θα έχει σαν αποτέλεσμα τα μέσα ενημέρωση αυτά για να κρατήσουν το κοινό τους, θα φροντίσουν αυτού του είδου το κοινό να είναι παρόν. Όταν κοιτάμε τηλεόραση, ε, ουσιαστικά κατοπτρίζεται ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Αν λοιπόν θέλουν πιο πολύ τα παραδοσιακά μέσα, πιο μεγάλη στην ηλικία από ότι νέοι, αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα στοιχείο που θα βοηθήσει στην εξέλιξη προς την σωστή κατεύθυνση. Και όταν μιλάτε για τη σεξιστική ρητορική των δημοσιογράφων ε, και ότι δεν είναι σύμμαχοι, δεν ήταν αυτό που θέλω να πω. Οι πληροφορίες που μας δίνονται, που παράγονται από τους δημοσιογράφους, πρέπει να συνάδουν περισσότερο στις προδιαγραφές ισότητας και ποικιλομορφίας. Και αυτό δεν θα έρθει απ' έξω. Θα έρθει και απ' έξω βέβαια και από την πίεση απ' έξω και πρέπει να πιέζουμε. Αλλά νομίζω ότι όσο οι ίδιοι επαγγελματίες δεν το συνειδητοποιούν, τότε θα προχωρήσουμε πάρα πολύ αργά. Ενώ αν μπορεί βέβαια να είναι ευσεβής πόθη, αλλά αν στις διάφορους ε, δημοσιογραφικούς οργανισμούς υπάρχει μια πολιτική ισότητας και επικοινομορφίας, μπορούν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι να συνδυτοποιήσουν και τότε τα πράγματα θα πάνε πιο γρήγορα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι σύμμαχοί μας οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί. Έτσι θα μπορούμε να έχουμε και μια ενημέρωση που να αντικατοπτρίζει πολύ περισσότερο την κατάσταση στην κοινωνία μας. Γιατί όταν φεύγουν από τη μέση οι γυναίκες ως δημοσιογράφοι, ε, τότε προφανώς και η άποψή τους εξαφανίζεται από την πληροφόρηση που φτάνει σε μας. Οι δημοσιογράφοι νομίζω ότι είναι έτοιμοι να το ακούσουν. Τώρα βέβαια οι συνθήκες εργασίας είναι τέτοιες που πολύ συχνά για να πάμε γρήγορα προσφεύγουμε σε στερεότυπα, τα οποία μας βοηθάνε να πάμε πιο γρήγορα. Ή προσφεύγουμε στον άντρα που θα είναι πάντα διαθέσιμος και σε 30 δευτερόλεπτα θα μας δώσει την πληροφορία που θέλουμε. Και αν έχουμε τρία θέματα να αναλύσουμε, δεν έχουμε καιρό να ψάξουμε να βρούμε τους σωστούς εμπειρογνώμονες, βρίσκουμε τον πρώτο διαθέσιμο. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα της ισότητας των φίλων συνδέεται με τον τρόπο που παράγεται η είδηση. Σήμερα οι δημοσιογράφοι υποβάλλονται σε τεράστιες πιέσεις. Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα και με μεγάλη βεβαιότητα όσον αφορά τη σταδιοδρομία τους να παράγουν την πληροφορία. Έχουμε το διαδίκτυο 24 ώρες το 24ωρο, οπότε όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και λαμβάνοντας τα υπόψη να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει η κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα, υπάρχουν και χρήστες και γυναίκες που είναι ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και το λένε, το φωνάζουν και είναι και ακριβώ τα κοινωνικά δίκτυα που μας επιτρέπουν να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να αφισβητήσουμε μια είδηση, μια πληροφορία Αμφισβητούμε λοιπόν κάποια είδηση, περιμένουμε να ζητήσουν συγγνώμη αυτοί που έφτεξαν. Οπότε η αντίδραση του κοινού και οι οργανώσεις γυναικών και φεμινιστών είναι κάτι που βοηθάει να λειτουργήσει καλύτερα η αυτορύθμιση και πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ θερμά. εγκάρδες ευχαριστήσεις προς τις τρεις εμπειρογνώμονες μας ε, που μας παρουσίασαν το θέμα από διαφορετική σκοπιά, επιστημονική, πανεπιστημιακή, ακτιβιστική, επαγγελματική. Ήταν πολύ χρήσιμες ε, οι παρατηρήσεις σας και θα αξιοποιηθούν δεόντως και στην εκπόνηση της έκθεσής μας. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα διακόψω μέχρι τις 5. Έχετε μισή ώρα διάλειμμα λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Περνάμε στο πέμπτο σημείο της ημέρησης διάταξης, το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοσιονομική Χρήση 2018. Όλα τα τμήματα. Συντάκτρια γνωμοδότηση τη Επιτροπή Γυναικών είναι η Μπάρμπαρα Ματέρα, αρμόδια καθήλυνα επιτροπή. Φυσικά, Επιτροπή Προπολογισμών. Γενικό Συγητή είναι ο κύριο Ζίκφρυντ Μουρεσάν, που έχει την καλοσύνη να έρθει στην Επιτροπή μα για να συζητήσουμε το θέμα. Θα του δώσω το λόγο για να μας κάνει την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσή του. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σα. Σας ευχαριστώ θερμά που με φιλοξενείτε σήμερα στην Επιτροπή σα. Ήρθελα από την έναρξη τη δημοσιονομική διαδικασία να μεταβώ σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές για να συζητήσουμε τους συναδέλφους τις προτεραιότητές μας για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Ε, μάλιστα, το Φεβρουάριο σας παρουσίασα το σχέδιο έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, το σχέδιο έκθεσης για τις κατευθυντήρες γραμμές για το προϋπολογισμό του 2018, με απαριθμίση των πολιτικών προτεραιοτήτων μας για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, το ψηφίσαμε τέλη Φεβρουαρίου και το Μάρτιο ψηφίσαμε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου με αρκετά μεγάλη πλειοψηφία έτσι έχουμε τις βασικές προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2018. Τώρα είμαστε στην επόμενη φάση. Είπαμε ότι δύο είναι οι πρωταρχικές μας προτεραιότητες. Η πρώτη ανάπτυξη και απασχόληση και δεύτερον ασφάλεια και προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί αυτές είναι οι προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών από εμά τώρα. Ανάπτυξη, οικονομική, απασχόληση, ασφάλεια και προστασία. Πώς θα υλοποιήσουμε τις προτεραιότητες. Ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση, καλό θα ήταν να επενδύσουμε σε τομεί που θα ενισχύσουν την οικονομία μας, θα την καταστήσουν πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική στις κρίσεις και άρα πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία, στις υποδομές, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην νεολαία, στο πρόγραμμα έρασμο, γιατί ο έρασμο δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα που εθαρρύνει του φοιτητέ να ταξιδέψουν, Άρα θα πρέπει να δείξουμε ότι ως φοιτητή αν έχεις ε, διεθνή πείρα Εμπλουτίζει το βιογραφικό σου και μπορεί να βρει πιο εύκολα δουλειά. 64% των εργοδοτών εκτιμούν ιδιαίτερα στην διεθνή πείρα στι προσλήψει που κάνουν. Οπότε θα πρέπει να ενισχύσουμε το έρασμος που αυξάνει την κινητικότητα των φοιτητών και καθιστά πιο ανταγωνιστικό το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη. Τέλη Μαρτίου λοιπόν υιοθετήσαμε τι κατευθυντήριε γραμμέ και το Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο προπολογισμού με βάση τι δικέ μα κατευθυντήριε γραμμέ. Μάλιστα, οι κατευθυντήριε γραμμέ μα σε μεγάλο βαθμό ελήφθησαν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότειναν το συν 7% δηλαδή για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την καινοτομία, γιατί όπως είπα, οι επενδύσεις στην καινοτομία και τις υποδομές θα έχουν κέρια σημασία για την ενίσχυση της οικονομίας. Συν 7% λοιπόν για το Ορίζοντα 2020, συν 8% για το Συνδέοντα στην Ευρώπη και συν 9% για το πρόγραμμα Έρασμος. Για το κόσμο, το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρότειναν μείον 2,6%. Θα το εξετάσουμε, γιατί σε σχέση με με πέρυσι το εξετάζουμε. Πέρυσι ήταν υπερβολικά αφύσικα υψηλό το ποσοστό, γι' αυτό και το μείωσε κάπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά θα το ελέγξουμε, γιατί δεν μπορούμε από τη μια να λέμε είναι προτεραιότητά μα οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και να περικόπτουμε τον περσινό προπολογισμό κατά 2,6%. Παρόλο που ο περσινό ήταν υπερβολικά διαγκωμένο. Πάντω το αρνητικό πρόσημο δεν είναι θετικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα επισκέφθηκα πολλές επιτροπές και διαπίστωσα την ετοιμότητά τους για τις υπο... επενδύσεις, ε, καινοτομία, υποδομές, ε, την ετοιμότητά τους να δώσουν προτεραιότητα στην καινοτομία στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες, στην υποστήριξη των μικρομεσαίων που δραστηριοποιούνται, δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Και μάλιστα Υπάρχει ανωδική τέτοια τάση, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού. Εμείς ε, σε αντίδραση θα είμαστε πιο φιλόδοξοι. Το επισήμαναν πολλοί συνάδελφοι στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ό,τι αφορά τη δεύτερη προτεραιότητα, την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών μας, θα πρέπει να φροντίσουμε οι διαθέσιμοι πόροι στις ε, γραμμές 3 και 4, που είναι περιορισμένες γιατί τις ε, χρησιμοποίησαμε πολύ εκτεταμένα στα, την προηγούμενη τελευταία διετία για να ξεπεράσουμε τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, διερωτήθηκα με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, πώς θα τους αξιοποιήσουμε. Χάρη στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών. Ζητήσαμε ενίσχυση της Europol, του Eurojust, Frontex, EASO ε, και ULIS. Αυτό κάναμε στην πρόταση. Φυσικά χρειάζεται αύξηση προπολογισμού και προσωπικού των σχετικών οργανισμών. Πρότεινε κάποιε αυξήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι ε, εφάμιλο όμως με τις προσδοκίε των οργανισμών. Θα δούμε λοιπόν ποιο είναι το σωστό ποσοστό αύξηση ε, στους προπολογισμού των οργανισμών. Πάντως είμαστε υπέρ ε, περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της άμυνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκεί που τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα και ακολουθεί και η βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα το κάνουμε. Με πρωταρχικό στόχο την εξοικονόμηση για να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος. Δεν μπορούμε να έχουμε 28 διαφορετικούς προϋπολογισμούς άμυνας ε, στις 28 χώρες μέλη για παρόμοια ή ίδια αποτελέσματα, εκεί που μπορούμε να κάνουμε οικονομίες και να έχουμε μία φορά αμυντικές δαπάνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να δρέψουμε από κοινού τους καρπούς. Επίσης, ε, θα έχουμε ασφάλεια στην Ευρώπη όταν ε, έχουμε ασφαλείς ε, γειτονικές χώρες. Γι' αυτό εμπλέκουμε στη συνεργασία της χώρες Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε της μετανάστευσης που πολλές φορές είναι η έλλειψη ευκαιριών σε πολλούς τομείς, διατροφή, υγεία, παιδεία, ακόμη και λόγω του κλίματος, ε, πόλεμοι. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της μετανάστευσης. Οπότε η Επιτροπή Προπολογισμών ανταποκρίνεται εν γέννη προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έμειναν όμως κάποιες εκκρεμότητες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, το, ε, ε, έχουμε 700 εκατομμύρια αποθεματικό στη Γεωργία. Γεωργικός προπολογισμό. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις κρίσεις. Έχουμε 332 εκατομμύρια αποθεματικό ε, για να συνεχιστεί ενδεχομένω ο μηχανισμό για του πρόσφυγε ε, σε, σχέση με, σε συνεργασία με την Τουρκία. Προ το παρόν δεν έχουν ε, προσημειωθεί κονδύλια. Έμεινε ένα περιθώριο. Θα δούμε αν υπάρχει πολιτική βούληση για τη συνέχιση αυτή τη πρωτοβουλία. Αν χρειαστούν, έχουμε μέχρι 232 εκατομμύρια. Αν χρειαστούν περισσότερα, θα πρέπει να τα βρούμε από αλλού. Και επίσης, επευκαιρία να δώσουμε και ένα μήνυμα επί της αρχής. Στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κυρίως απέναντι στο Συμβούλιο, θα πούμε με σαφήνεια ότι αν περιμένουμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες, θα χρειαστούμε και φρέσκο χρήμα, νέα κονδύλια. Δεν θέλουμε να διακυβεύσουμε υφιστάμενα προγράμματα που ήδη τρέχουν. Αν θέλουμε νέες προτεραιότητες και νέες αρμοδιότητες, χρειάζονται και νέοι οικονομικοί και δημοσιονομικοί πόροι. Γιατί δεν θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να υπονομευθούν τα τρέχοντα προγράμματα. Το Μάρτιο στις κατευθυντήριες γραμμές, κυρία Πρόεδρε, και φτάνω στο τέλος ε, της παρέμβασης, περιλάβαμε και τη συνεκτίμηση του φίλου όπου είναι δυνατό στις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το περιέλαβα και στις κατευθυντήριες γραμμές του Μαρτίου. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες δικής Επιτροπής για το 2018, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ε, αυξάνεται κατά 1,2% το πρόγραμμα για τα δικαιώματα, ισότητα και την ηθαγένεια ε, για τη σχετική δημοσιονομική γραμμή που προωθεί την πάταξη των ε, ε, διακρίσεων αυξάνεται κατά 2%. Υπάρχει αύξηση ό,τι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων. Έχουμε περισσότερες υποχρεώσεις από ό,τι πέρυσι και έχουμε αύξηση και στις πληρωμές. Οπότε θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ε, δράσεις στους δικαιούχους και του χρόνου και έχουμε αύξηση 4,6% σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις μεταπληρωμών από την περασμένη φορά. Ελπίζω να μείνατε ικανοποιημένοι με αυτές τις ε, αυξήσεις. Πείτε μας αν θεωρείτε ότι είναι ανεπαρκής και αυτό θα γίνει συζήτηση μετά και η γνώμη σας μετράει. Για να ενισχυθεί πάντως η διαφάνεια και η καλύτερη προβολή, η ορατότητα των ταμείων, των κονδυλίων, Ίσως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια νέα γραμμή στο πρόγραμμα, ώστε να υλοποιήσουμε ακριβώ αυτό το στόχο τη εξασφάλιση διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, στο σχέδιο προπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το ίδιο προσωπικό, χωρί αύξηση του προσωπικού σε σχέση με πέρυσι, ούτε αύξηση ούτε μείωση. Κάτι που ευθυγραμμίζεται και με τα αιτήματα του οργανισμού. Αυτό ζήτησε ο οργανισμό να συνεχιστεί ε, το ίδιο επίπεδο υπαλλήλων. Είπαν λοιπόν, ότι δεν χρειάζονται επιπλέον προσωπικό, αλλά ούτε φυσικά ε, είναι σκόπιμη η μείωση του προσωπικού. Εσείς τι γνώμη έχετε. Πιστεύετε ότι χρειάζεται περικοπή ή αύξηση. Περιμένω και τις δικές σας προτάσεις. Πάντως ε, για τον οργανισμό γενικώ αυξάνεται κατά 2,1% ο 2,1% αυξάνεται ο προπολογισμό του οργανισμού συνολικά, αλλά το προσωπικό μένει το ίδιο με πέρυσι. Επίσης, ε, τα επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο ξεκίνησαν με πολύ αργούς ρυθμούς κατά την αρχή του πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου και η διαπίστευση των αρχών διαχείρισης επίσης καθυστέρησε. Τώρα αρχίζουμε και αποκτούμε κάποιο ρυθμό κουραζιέρας. 469 από τις 564 αρχές έχουν αρχίσει και λειτουργούν, εθνικές αρχές, οπότε μπορούμε πια να προβαίνουμε σε πληρωμές. Και από τη, και από τη στιγμή που συντρέχουν οι, προθέσεις, οι προϋποθέσεις σε εθνικό επίπεδο για να γίνουν πληρωμές, περιμένουμε το χρόνο αύξηση των αιτήσεων. Οπότε με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που σας ενδιαφέρει, τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, ήδη έχουν τις συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση στις πληρωμές, στα κονδύλια. Και στο 1β, στο 1β κεφάλαιο, ε, διαρθρωτικά και ταμείο συνοχή, ζητήσαμε αύξηση του επίπεδου πληρωμών. Μέχρι στιγμή δεν χρειαζόταν τόσε πολλέ πληρωμέ, γιατί δεν υπήρχαν δομέ και δεν υπήρχαν αιτήματα από τα κράτη-μέλη. Από τη στιγμή που έχουν εξασφαλιστεί υποδομέ, από το χρόνο θα ενισχυθεί ο ρυθμός απορρόφησης των κρατών μελών. Οπότε θα πρέπει να έχουμε περισσότερες, ε, περισσότερα κονδύλια πιστώσεις πληρωμών στον τομέα 1β. Γιατί το χειρότερο μήνυμα που θα μπορούσαμε να δώσουμε στο κοινό είναι ότι δεν είμαστε σε θέση να πληρώνουμε τους, οργαν... τους λογαριασμούς μας, τα χρωστούμενα και να... να πληρώνουμε τους δικαιούχους. Γι' αυτό και προτείναμε αύξηση των πιστώσεων πληρωμών στο τομέα 1β. Δεν ξέρω αν το θεωρείτε επαρκές το ποσοστό αύξηση που προτείνουμε. Αυτά και η σημερινή μου παρουσία είναι απλώς η αρχή του διαλόγου και της συνεργασίας μας. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, να έχετε υπόψη ότι θα ψηφίσουμε το σχέδιο έκθεσης ε, για την εντολή για τον θερινό τριμερή διάλογο, δηλαδή για να Υποβάλλουμε στο Συμβούλιο και την ε, Επιτροπή το, την πρόταση που σας παρουσίασα, θα ψηφίσουμε στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια για την εντολή για να δει το Συμβούλιο και η Επιτροπή ποιες είναι οι προτεραιότητες μας και πού βρισκόμαστε. Το πιο σημαντικό βέβαια θα είναι οι φθινοπορεινές διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό και λέω ότι τώρα είναι η έναρξη της συνεργασίας μας. Και μην διστάσετε στους επόμενους μήνες να έρθετε να με βρείτε και να μου επισημάνετε σημεία που κατά τη γνώμη σας είναι σημαντικά, γιατί όσο περισσότερα επιχείρηματα έχω, τόσο καλύτερα θα προσπίσω τις κοινέ μας προτεραιότητες, τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, ε, με την Επιτροπή και κυρίως με το Συμβούλιο. Και το Συμβούλιο είναι που επιχειρεί πολύ τακτικά να επιβάλλει περικοπές στα κονδύλια του προπολογισμού. Οπότε όσο περισσότερα επιχειρήματα ε, θα συνηγορήσουν υπέρ των προτεραιοτήτων μας τόσο το καλύτερο. Τα περιμένω. Αυτά και περιμένω συνεργασία και διάλογο και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μουρασάν. Ας ακούσουμε τώρα και τους συναδέλφους της Επιτροπής μας. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Ματέρα που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Μου έστειλε όμως το εξής μήνυμα που με χαρά θα σας διαβάσω εκ μέρους της. Είναι χαρά, μας λέει η κυρία Ματέρα, που καλωσορίζουμε τον κύριο Μουρεσάν, ε, εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό. Οι δραστηριότητες πρέπει να εξυπηρετούν στους μακροπρόθεσμους στόχους, επαρκείς δηλαδή χρηματοδοτήσεις για τα θέματα του προγράμματος Δάφνε για την ε, ισότητα και για την ανάπτυξη της γυναίκας, ε, κοινωνικά και οικονομικά θέματα στην ψηφιακή οικονομία, στον τομέα της ε, κοινωνίας πληροφορίας, συμμετοχή των γυναικών στις επιστήμες, όπου, στον επιστημονικό κόσμο που είναι σημαντικό το χάσμα ακόμη μεταξύ ανδρών και γυναικών, προκειμένου να ε, επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι πρέπει η ενσωμάτωση θέση του φύλου να μπει και στο δημοσιονομικό σχεδιασμό που πρέπει να καταστρέψει εκ τούτου εργαλείο χρήσιμο για την προαγωγή της όδο μεταξύ ανδρών και γυναικών σε μια ευρύτερη προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να καταστήσουμε την ε, ενσωμάτωση της του φύλου στον προϋπολογισμό ως πυλώνα του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και στι προσεχεί λοιπόν δημοσιονομικέ προεπτικέ πρέπει να προβλεφθεί ειδική γραμμή για τον προπολογισμό με ενίσχυση των πόρων για του ειδικού στόχου του προγράμματο Δάφνη. Επίση, πολύ σημαντικό, δύο σημεία ιδιαίτερα. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπως το ορίζουν 2020 και τα κοινωνικά ταμεία πρέπει να προβάλλουν ιδιαίτερα τις γυναίκες στο χώρο της επιχειρηματικότητας, πρόσβαση στα δάνεια, και χρηματοδότηση για επιχειρηματικές δραστηριότητες και η καταπολέμηση της βίας φάρας των γυναικών πρέπει να ε, προωθηθεί από το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων με την ε, πραγματογνωμοσύνη και τους πόρους που θα πρέπει να τεθούν ώστε να απαφευχθούν επικίνδυνες ε, και περιττές επαναλήψεις δράσεως ή επικαλύψεις μεταξύ των υπηρεσιών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ενίσχυση της διάστασης των φύλων για την επιτεύξη των δοχών αυτών και ελπίζω ο εισηγητής κ. Μόρεσαν να εστερνιστεί τις απόψεις μας. Αυτό ήταν το μήνυμα της ε, συντάκτης της ομοδοτήσεώς μας, κυρίας Ματέρα. Και τώρα θα παρακαλέσω τους κοιόδες μας να λάβουν το λόγο με την κυρία Μούντι πρώτα εκ μέρους των Δημοκρατών. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή των Γυναικών των δικαιωμάτων των γυναικών. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στα όσα ήδη επισημάνθηκαν από την κυρία Ματέρα, ερήμην για την έκθεση αυτή. Ιδιαίτερος η ιδέα της ενσωμάτωσης του φίλου στο δημοσιονομικό σχεδιασμό και πάνω απ' όλα η ανάγκη να μην λησμονούμε την τάσταση του φύλου και όλη την προστιθέμενη αξία ε, που μπορεί να εξασφαλίσει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στο θέμα αυτό με την αναγκαία αναγνώριση της ανάγκης για προαγωγή μιας από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της ισότητας των φύλων. Ταυτόχρονα όμως και στο σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη. Το μιλούμε για τις ε, υποδομές. Συχνά γίνεται λόγος μόνο για γέφυρες, δρόμους, αεροδρόμια, αλλά πρέπει και τις κοινωνικές υποδομές να ενισχύσουμε. Η οικονομική ανάπτυξη αποδεικνύεται πολύ πιο αποτελεσματική όταν ενισχύεται και η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα. Πολύ περισσότερο από ότι τα υλικά αυτά έργα, τα κατασκευαστικά αυτά έργα των υποδομών που ανέφερα. Καλωσορίζω και πάλι λοιπόν τα σχόλια που ακούστηκαν, ιδιαίτερα για το πρόγραμμα Δάφνη, για τα δικαιώματα, την ισότητα, τη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών και επίσης ε, στη χρηματοδότηση, το έτσε αλλά και τα λοιπά ταμεία για τα οποία έχει γίνει λόγος. Και ξέρω βεβαίως ότι υπάρχει το ζήτημα ή το ζητούμενο καλύτερα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά γενικότερα το θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου στα ταμεία αυτά, που ε, συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δίνουν λόγο τα ταμεία και για τον αντίκτυπο των δρασεών τους ε, στο θεματολόγιο το σχετικό με την ισότιμη αντιμετώπιση των φύλων. Και βέβαια όλα αυτά συμπληρωματικά στα όσα είπε η κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ η κυρία Χάνιμπολ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα συμφωνήσω βέβαια και με την Κλερμούντι και με την Μπάρμπαρα Ματέρα μια όμως και είστε εδώ, δράτω με τις ευκαιρίες, αν το επιτρέπουν οι συνάδελφοι της Επιτροπής, να μιλήσω και για την ε, ασφάλεια και τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Εγώ ε, εκπροσωπώ την εκλογική περιφέρεια του Λονδίνου. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας περιγράψω τι αισθάνεται κανείς όταν ξυπνάει το πρωί μιας Κυριακής για να διαπιστώσει ότι λίγο πιο κάτω στον δρόμο που μένει έχει σκάσει μια βόμβα. Είναι κάτι που βλέπουμε στην Βρετανία αλλά όχι μόνο στη Βρετανία. Δεν αφορά μόνο το Λονδίνο, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Βέβαια στο Λονδίνο είχαμε δύο τρομοκρατικέ επιθέσει, αλλά και εκείνη του Μάντσεστερ τι τελευταίε εβδομάδε. Αλλά είχαμε και μεγάλε επιθέσει και στι Βρυξέλλε και στο Παρίσι. Άρα καθίσατε τρομοκρατία και η ασφάλεια όλο και πιο ευρωπαϊκού χαρακτήρα και διάσταση θέμα. Χαίρομαι για τα όσα είπατε και χαίρομαι που η Επιτροπή των Προπολογισμών λαμβάνει υπόψη τι ε, παρατηρήσει αυτέ. Η ενίσχυση των υπηρεσιών όπω τη Europol και τη Eurojustice βεβαίω είναι εξαιρετική εξαιρετική ιδέα, πάρα πολύ καλή ιδέα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το συλλογισμό και να κοιτάξουμε περισσότερο πώς μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον κάποιες από τις ρίζες της τρομοκρατίας. Γιατί κάποιοι αισθάνονται ότι πρέπει να καταφύγουν στην τρομοκρατία. Και εδώ έχει το ρόλο της και η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, αλλά ιδιαίτερα και η κοινωνική συνοχή. Αυτά που προσφέρει δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο, όπως και άλλα ταμεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα και ξέρω ότι είναι προτεραιότητά σα βέβαια η ασφαλεία και η καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Ε, όμως ιδιαίτερα πρέπει σε αυτό να σταθούμε και να δώσουμε κύρια προτεραιότητα γιατί είναι και το κύριο μέλημα η περιπτώσει είναι πρώτο στα μελήματα των Ευρωπαίων πολιτών το θέμα τη Τρομοκρατία, σε ορισμένε χώρε περισσότερο από κάτι, κάποια άλλη. Αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνο και η ανησυχία ότι μπορεί να διαχυθεί το φαινόμενο από τη μία χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην άλλη και πρέπει να του δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Ευχαριστώ κύριο Σαρτασούν. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μωρισάν που ήρθατε σήμερα. Σας ευχαριστώ και που είσαστε έτοιμος να συνεργαστείτε και να ακούσετε τις διάφορες κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Θέλω όμως να επιμείνω στο θέμα του προπολογισμού για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων δεν ε, υπάρχει, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και θα έπρεπε να διορθωθεί. Για να βγούμε από την κρίση, είναι πολύ σημαντικό το πού θα επενδύσουμε, πού θα κατευθύνουμε τις επενδύσεις. Και από αυτό θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα αποφελθούν και οι άντρες και οι γυναίκες ή όχι. Χάρηκα που άκουσα ότι ο προπολογισμό του Ινστιτούτου θα αυξηθεί. Είναι κάτι που ενδιαφέρει την Επιτροπή μας. Εγώ προσωπικά έχω συνεργαστεί πολύ καλά. Νομίζω ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και πρέπει να στηρίξουμε τις δραστηριότητές τους Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πολλές και χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, ε, για δικαιώματα των γυναικών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε τον κανόνα της κυβέρνησης Τραμπ να μην υποστηρίζει πια μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα της υγείας και των ε, αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάτι για να στηρίξουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αυτές, στις οποίες αποφάσισε να κόψει τη χρηματοδότηση ο πρόεδρος Τραμπ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι ειδικό επί του προϋπολογισμού, λέει ο κύριος Μαρτά. Θέλω να συγχαρώ τους διερμηνείς, λέει ο μιλητής, γιατί μιλούσατε πάρα πολύ γρήγορα και μπράβο που τα κατάφεραν. Το να μιλάμε για την ε, καινοτομία είναι φυσικά κάτι με το οποίο συμφωνώ κι εγώ. Συζητάμε νομοθετικές εκθέσεις για την ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή ένωση κλπ. Και Υπάρχει όμως και τάση που δεν πάει εκεί. Να δούμε λοιπόν πώς θα τα βάλουμε αυτά μαζί. Μερικές φορές ψηφίζουμε κάποια πράγματα, αλλά ο προπολογισμό έχει άλλες προτεραιότητες. Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερον, αν κατάλαβα καλά, το λέω θετικά έτσι, μιλήσατε για πάνω από 25% της 1αβ, δεν έχει σημασία, είναι αλήθεια, όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν δομές, υποδομές που θα έπρεπε να υποφελούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, διαμαρτύρονται όμως γιατί οι πληρωμές γίνονται με τεράστια καθυστέρηση, κάτι το οποίο τους δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες. Όταν ζητάει κάποιος χρηματοδότηση, αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο, δύσκολο και αν επιπλέον έχει να υποστεί και καθυστερήσει στις πληρωμές, ίσα καταλαβαίνετε ότι τις βάζει σε τεράστια δυσκολία και από αυτού λοιπόν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα. Παρακαλώ, κύριε Μούρισαν τα συμπεράσματά σας, οι απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συναδελφοί, για όλα τα στοιχεία που μου δώσατε. Κύριε Μαρτά, ναι, έχετε δίκιο για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Υπάρχουν ήταν πραγματικότητα και στο παρελθόν, κυρίως γιατί στο προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο πολύ συχνά οι χώρες μέλη στη δεύτερη κολόνα με τις πληρωμές θέλουν να κρατήσουν το επίπεδο όσο γίνεται πιο χαμηλό. Πράγμα που σημαίνει ότι τα rest αλικητέ, τα καθυστερημένα δηλαδή, συσσωρεύτηκαν από την προηγούμενη περίοδο και φτάσαμε το 2015 και 2016 και καταφέραμε τότε να πληρώσουμε ε, τις οφειλές αυτές, τους λογαριασμούς αυτούς τους απλήρωτους. Στην αρχή της περίοδου είναι πάντα ε, μικρή η καθυστέρηση, αλλά σίγουρα αυτή τη φορά πρέπει να προσπαθήσουμε σε αυτή την περίοδο να μην καταλήξουμε στα ίδια. Δηλαδή όταν οι χώρες μέλη απορροφούν κονδύλια θα πρέπει να στέλνουν τους λογαριασμούς και να ξέρουμε από την αρχή Είπαμε 25% συν πληρωμές πρέπει να φροντίσουμε τις επόμενες χρονιές να πληρώνουμε. Έχετε δίκιο όμω και για την γραφειοκρατία. Είναι ένα εμπόδιο όχι τόσο για τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο για τις μικρές. Οι τεράστιε ε, αρχιοθετούν ε, έγγραφα, συμπληρώνουν, έχουν δικηγόρου, λογιστές κτλ. Αλλά άλλοι, οι νέοι επιχειρηματίες που έχουν μια μικρή επιχείρηση, αν πρέπει για πέντε χρόνια να αρχιοθετήσουν ένα έγγραφο, να συμπληρώσουν δεν ξέρω άλλα, αυτό είναι τεράστιο γραφειοκρατικό άκθος, το οποίο τους οδηγεί μερικές φορές και σε αποτυχία. Αυτό πρέπει να απλοποιηθεί λοιπόν, έχετε δίκιο και το κάνουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών με μελέτες για το κόστος της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πόσο κοστίζει για ένα ευρώ, πόσο κοστίζει στον δικαιούχο. Για τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και για τον κίνδυνο το ότι μπορεί να χρειαστείς ε, κάποιους συμβούλους για να προετοιμάσεις το φάκελό χωρίς να είσαι καν σίγουρος ότι θα επιλεχθείς και θα, θα χρηματοδοτηθείς. Το έχουμε υπόψη μας αυτό και θα φροντίσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών να το φροντίσουμε. Το σημείωσα και αυτά που είπε κλωτμούδη και ο κ. Σορτασούν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικικών Επενδύσεων. Ξέρετε, θα έπρεπε να γίνονται καλύτεροι υπολογισμοί και να μην υπάρχει διάκριση σε βάρος των γυναικών που ζητούν χρηματοδότηση. Τα ίδια και για τις κοινωνικές υποδομές. Έχετε δίκιο και το σημειώνουμε. Ασφάλεια επίσης. Ένας από τους λόγους για τον οποίο πιέζονται οι επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη είναι να έχουμε καλύτερες πληροφορίες. Αν υπάρχουν κάποιες υπόνοιες για λαθροδιακίνηση, για τρομοκρατία, Χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια στα εξωτερικά μας σύνορα. Αν οι υπηρεσίες μας ενισχυθούν, τότε θα τα καταφέρουμε καλύτερα και αν συνεργαστούν καλύτερα μεταξύ τους. Αυτά νομίζω ότι ήταν τα κύρια σημεία για το Δάφνη και την πρόοδο ναι, από τη δικιά μου την πλευρά να λαμβάνω την υποχρέωση να φροντίσω για κατάλληλη χρηματοδότηση στον επόμενο προπολογισμό. Όπως είπα, στις διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σας χρειάζομαι, να ξέρω πώς αξιολογείτε την κατάσταση. Τι συμβαίνει με τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα τα πάρω μαζί μου. Δεν διαφωνώ με κανένα. Όλα είναι πολύ καλά σημεία. Και θα είμαι σε επαφή μαζί σας και θα συνεργαστούμε μαζί τους επόμενους μήνες εν ώψη του προπολογισμού. Ευχαριστώ και εμείς προσβλέπουμε σε πολύ αγαστή συνεργασία και ελπίζουμε επίσης ότι θα λάβετε εδώ υπόψη και τις δικές μας προτεραιότητες. Next point on Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης της που προβλέπει ψηφοφορίες. Έχουμε ε, το σημείο 6 της ημέρησης διάταξης. Είστε έτοιμοι, έχετε τις κάρτες, ψηφ... τις κάρτες ψηφοφορίας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε και ηλεκτρονικά χρειαστεί. Λοιπόν, το σημείο 6. το σχέδιο θέση με τη μορφή τροπολογιών με θέμα την καταπολέμηση των ανισοτήτων, ως μοχλό για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης. Η συντάκτρια, η συγκήτρια μάλλον της θέσης μας είναι η κυρία Γνιέσκα Κοζόφσκα Μαγιάννης. Ποιος είναι υπέρ για την τροπολογία 9 κατά, αποχές. Δυστυχώς πρέπει να το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά, οπότε άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 9, παρακαλώ. Δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Κατά τμήματα, σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 10. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται έτσι. Τροπολογία 26. Ποιος είναι, σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ε, υπάρχει και προφορική τροπολογία για αυτό το σημείο, για την τροπολογία 2. Μήπως υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Όχι. Οπότε θα ψηφίσουμε τα, κατα, τα κατατήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με την προφορική τροπολογία. ποιο είναι ή όχι. Ναι. Δεύτερο τμήμα με την προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται.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 Mm-hmm. Uh, now, we will vote on the report Ψηφίζουμε την έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της ε, σεξουαλικής εκμεταλλεύσης και ε, καταχρήσεως βάρος των παιδιών παιδική πορνογραφία. Ξεκινούμε την ψηφοφορία. Συμβαστική υπαριθμών 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε αλφα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 21, προφορικά, προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην προφορική τροπολογία. Την ψηφίζουμε λοιπόν. 21, με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. πέρασε Και εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 37 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στη 42 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 με προφορική τροπολογία της εισηγητρίας. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω μια προφορική τροπολογία στην προφορική τροπολογία. Το κείμενο που έχετε εσείς τώρα με την ε, πρώτη, τροπολογία, με την πρώτη προφορική τροπολογία θα συνεχίσει, αλλά θα βγει ο, η φράση «ταξιδεύουν στο εξωτερικό και επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και θα μείνουμε και θα συνεχιστεί από εκεί, μένει αυτό και συνεχίζεται στο for sexual purposes, δηλαδή βγαίνει για, για ε, αναψυχή, για διακοπές. Ε, υπάρχουν αντιρρήσεις, λέει η Πρόεδρος, όχι. Την 49 λοιπόν με την προφορική τροπολογία. 49 λοιπόν με προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, μάλλον με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Όχι, στο σύνολο. της τροπολογίας. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμόν 1 με προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις στην προφορική την υπαριθμόν 1 λοιπόν με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική υπαριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. Επτά. Προφόρικη τροπολογία. Αντιρρήσεις. Επτά, λοιπόν. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε παρακαλώ. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Και εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Καμία ψήφος κατά. Και πέντε αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Κλεριμούντι. Αγαπητοί συνάδελφοι, 12 Ιουλίου το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ και πέρα συνεδριά σας. Ah, uh, thank, you very much for, the interpreters and thank you very much. Η πρόεδρος ευχαριστεί τους διερμηνές και ευχαριστούμε πολύ και τη γραμματεία. Και εμείς ευχαριστούμε.